Να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν αρκετά μέλη εδώ, ποιοτικά μέλη, να ξεκινήσουμε τις ε, συζητήσεις. Καταρχάς, ζητώ αν εγκρίνετε, να πείτε αν εγκρίνετε τη μερίσια διάταξη. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα μπροστά σας, το εγκρίνετε. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, ή αν δεν θέλετε να θέσετε κάποια ζητήματα, προχωράμε και πάμε στην έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου. Και ξανά, αν δεν υπάρχουν σχόλια ή αλλαγές, θεωρούνται συμπεφωνημένα. Θα προβώ σε κάποιες ε, ανακοινώσεις εκ μέρους της Προέδρου. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αύριο 5η 21 Μαρτίου από τις 30 έχουμε αλλαγή αίθουσας συνεδρίασης. Στα, είμαστε στην PHS 3C050 απέναντι στην Πασαρέλα στις 9 η ώρα διότι θα διεξαχθεί οικονομικός διάλογος ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο τον καινούριο του κύριο Γκρόπ τον κύριο Μπλουέμ. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του. Και σημείο 9 για συνταγματικά προβλήματα για διακυβέρνηση πολυεπίπεδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγγήτρια κυρία Γκουλάρ, τα μέλη να γνωρίζουν ότι όσον αφορά συγκεκριμένο θέμα, οι τροπολογίε για τη γνωμοδότηση για τα συνταγματικά προβλήματα τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω ανεβλήθη για άλλη συνεδρίαση. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτό να το εξετάσουμε. Αυτέ είναι οι μόνε ανακοινώσει που πρέπει να κάνω. Και χωρί να χρονοτριβώ, πάμε στην ε, πρώτη έκθεση. Είναι εδώ η συγγήτρια η κυρία Μόνικα Κλίβα, που, Μόνικα Κλίβα θα παρουσιάσει λοιπόν τη γνωμοδότησή της σχετικά με την έκθεση που αφορά την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς, να πω στους συναδέλφους που έβαλαν 236 ε, τροπολογίες ότι τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους και όδους ηγητές όλους ιδιαίτερος με τους οποίους καταφέραμε να συναντηθούμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και να προβούμε σε πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτινόμενες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Εκτιμώ όλα τα σχόλια των ε, συναδέλφων και νομίζω ότι στο τέλος σημερινής ημέρας θα έχουμε ενημερωμένη εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών που θα τις στείλω στο τέλος της ημέρας, μέχρι το τέλος της ημέρας. Περιμένω να ακούσω τη συζήτηση για να διευκρινιστούν κάποιες τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες πριν επικαιροποιήσω τις ε, τροπολογίες. Το θέμα ε, τελικά αποκτά ορμή στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής και εν γέννη γίνεται επίκαιρο. Θα ήθελα η έκθεση να είναι στεναρή που θα δείχνει σαφώς τη θέση του Κοινοβουλίου και νομίζω με τις 26 συμβαστικές τροπολογίες κατευθυνόμαστε προς την ε, ορθή κατεύθυνση. Αυτή είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό μας επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση των απαιτήσεών μας και των ιδεών μας. Ε, Παρ' όλα αυτά θα ήθελα το Συμβούλιο όλος ιδιαίτερος να μας πάει στα σοβαρά και ελπίζω ότι θα πετύχουμε ισχυρή πλειοψηφία στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Μαΐου που θα υποστηρίξει εν σαφείς ορισμούς των φορολογικών παραδείσων και θα παρουσιαστεί μια σαφής γραμμή προτάσεων για επιβολή κυρώσεων όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Πολλές τροπολογίες ε, κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συζήτηση θα ακούσω περισσότερο τις απόψεις συναδέλφων των τροπολογιών, αλλά κάποια λεπτά, λεπτά θα ήθελα να αναφερθώ στην παρούσα πρόταση που έχω για τις συμβαστικέ. Με τα χαράς βλέπω ότι κάποιες τροπολογίες τονίζουν και υπογραμμίζουν τον ε, ρόλο των αυξανόμενα σημαντικό που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές προσκήνιο θα πρέπει τα συμπεράσματα αυτή τη εκθέσεω να τροφοδοτηθούν όχι μόνο προ του πολιτικού μα ηγέτε και τα θεσμικά όργανα, αλλά και προ τι συζητήσει του ΟΣΑ, των G20, του Global Forum και των G8. Ε, οι ευρωπαϊκές αρχές της διαφάνειας, αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και κατάργησης βλαβερών φορολογικών πρακτικών πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που θα μας καθοδηγούν όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και τις σχετικές διαδικασίες. Ε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά αυτό θα προτείνω ξεχωριστό κεφάλαιο στην έκθεση που θα καλύπτει και θα συγκεράζει όλες τις ιδέες που αφορούν τη φορολογική απάτη, τις φορολογικούς παραδείσους σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα το ονομάσω το κεφάλαιο αυτό Διεθνής Διάσταση. Εκεί θα συμπεριληφθούν τα σχετικά σημεία. Το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα αυτό στη συνεδρία των Σκιωδών, διότι υπήρχαν πολλέ ε, τροπολογίε Επιτροπή Ανάπτυξη και άρα αυτή είναι καλή λύση, πιστεύω. Επίση, με τα χαρά να συζητήσουμε περαιτέρω την ιδέα του να δώσουμε σε αρμόδιε αρχέ την εξουσία να αναλάβουν δράση και να αναστείλουν τις άδειες τις τρα, ε, τραπεζικές στους χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν διαπράττουν απάτες προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες ούτως ώστε να αποφύγουν τη φορολόγηση ή αρνούνται να συνεργαστούν με τις φορολογικές αρχές. Ήταν ένα από τα ισχυρά σημεία της έκθεσης και υπήρξαν σχετικές τροπολογίες. Έτυχε μεγάλη υποστήριξη αυτή η προσέγγιση και η έκθεση θα επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τη σχετική οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος που δημοσιεύθηκε ακριβώς όταν εμείς ετοιμάζαμε την έκθεση. Οπότε πολλές τροπολογίες ε, υπάρχουν για αυτό το σημείο που είναι κρισίμου σημασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνει την πρόταση εισάγοντας την υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν δημόσια μητρώα, κυβερνητικά που θα είναι διαθέσιμα όσον αφορά τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες και συμμετοχή σε διάφορες εταιρείε, καταπιστεύματα κλπ. Και, άλλους, και άλλα νομικά πρόσωπα που αυτό θυραμίζουν την έκθεση. Και τελικά καλωσορίζω και άλλες ιδέες των συναδέλφων σχετικά με τη συζήτηση ε, για την ε, τιμολόγηση των μεταφορών η μεταφορά των κερδών σε φορολογικού ε, παραδείσου από αναπτυσσόμενε χώρες χώρε για την αποφυγή φορολόγηση είναι ένα πρόβλημα που πετύχει άμεση δράση από πλευρά ευρωπαϊκή αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΩΣΑ όσον αφορά την τιμολόγηση των μεταφορών ποσών κονδυλίων αλλά και αναθεώρηση των υποχρέωσεων που υπάρχουν σύμφωνα με την νομοθεσία τη σχετική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την τιμολόγηση των μεταφορών και τι διάφορε κατευθυντήριε γραμμέ. Είναι κάτι που απαιτείται. Ευχαριστώ του Κιώδη και όλου όσου υπέβαλαν τροπολογίε σχετικά με την έκθεση. Προσβλέπω σε περαιτέρω σχόλια και βέβαια θέλουμε να έχουμε καλά εδρεωμένε συμβαστικέ προτάσει και θέλουμε μια ισχυρή έκθεση του Κοινοβουλίου αυτού του ζητήματο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> την εισηγήτρια. Οι πολιτικές ομάδες τώρα. Η κυρία Πιετικά είναι για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και τους άλλους κοιόδης εισηγητέ για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για τις συμβαστικές λύσεις μπορώ να υποστηρίξω την κοινή γραμμή που αναλάβαμε για τον καθορισμό, για τους καθορισμούς, για να έχουμε και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών στις διάφορες χώρες. και τις ε, κοινέ ε, αντιμετωπίσεις των φορολογικών αδικημάτων και κυρίως τα δικήματα που συνάπτονται με τα προβλήματα αυτά αναφέρονται στην οδηγία κατά, της, κατά του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος για τους φορολογικούς παραδείσους πρέπει να υπάρξει σαφήνεια και εδώ βασιζόμαστε σε διεθνούς χαρακτήρα ορισμούς που μπορούμε να έχουμε για την έννοια του φορολογικού παραδείσου Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια σωστή εξισορρόπηση εξουσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα ίδια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε ακόμα καλύτερα την ε, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπογραμμιστούν όλες αυτές οι ιδέες και εάν συμφωνείτε και οι υπόλοιποι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να έχουμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου για τα θέματα φορολογικής απάτης και επιθετικής κατά κάποιο τρόπο σχεδίασης για την αποφυγή φόρων. Γιατί αυτά αξίζουν μια πλήρη συζήτηση. Κάποιες ιδέες που θέλω επίσης να υπογραμμίσω. Θα ήθελα να έχουμε μεγάλη σαφήνεια και να είμαστε συγκεκριμένοι στα θέματα διεθνούς χαρακτήρα να μπορέσουμε να παροτρύνουμε όλους να προχωρήσουν σε μια συμφωνία στα πλαίσια του ΟΣΑ για αυτόματη ε, ανταλλαγή πληροφοριών από τους υπευθύνους στα, διάφορα κράτη-μέλη του ΟΣΑ και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε σαφήνεια γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να δίνουν οποιαδήποτε επιδότηση ή πρόσβαση σε δημοσίους διαγωνισμούς σε οποιοδήποτε φορέα επιχείρηση που έχει καταδειχθεί ότι εμπλέκεται σε οικονομικά δικήματα. Για την τιμολόγηση εκμεταφοράς έχουμε ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε εδώ. Η πρόκειται για τις συμφωνίες για τιμολόγηση εκ των προτέρων και αυτό μπορεί να είναι ένα αντίμετρο στην εκμεταφορά στη τιμολόγηση και επομένως η αποφυγή αυτή τη πρακτική θα πρέπει να προσθεθεί στις κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως για κάθε συναλλαγή θα πρέπει να καταγράφεται η καταρχήν τιμολόγηση και οι επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με φορολογικούς παραδείσους θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση και τον προορισμό των χρημάτων που προκύπτουν από την συναλλαγή και για τους επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η συναλλαγή και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να υπάρξει και μια περιορισμένη αναθεώρηση για την οδηγία περιλογιστικής καταγραφής ώστε να υπάρχει μια χωριστή καταγραφή της ε, εταιρείας συμμετοχών, των εταιριών συμμετοχών για τα θέματα αυτά. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στα εργαλεία, μετά θα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και επίσης θα ασκηθεί και δημόσια πίεση εναντίον των φορέων αυτών που παραβιάσουν τους κανόνες. Ευχαριστώ. Okay. Uh, and... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άικου, εκ μέρους των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι η άλλη δεν είχε το λόγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι εδώ Πρόεδρε, κανένα πρόβλημα δεν έχω, ούτε φέρω αντίρρηση στο πρόγραμμά σα. Ευχαριστώ λοιπόν και την εισηγήτρια για την έκθεση και μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων για τι συμβαστικέ τροπολογίε Θα είμαι εξαιρετικά σύντομο, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να εξεύρουμε κάποιον, ε, κάποια ισορροπία και ένα συμβιβασμό μεταξύ των ε, ομάδων στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ε, για το ζήτημα αυτό των φορολογικών παραδείσων, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ε, όλοι σχεδόν ε, συμφωνήσαμε, σχεδόν όλοι, σίγουρα θα παρέμετε στη συνέχεια, συνάδελφε. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε βρει αυτή την ισορροπία που θέλαμε μεταξύ των ομάδων. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είμαι Ολλανδός. Γνωρίζω ότι η κυβέρνησή μου θα ήθελε να αποφύγει ε, να υπάγεται και δική μου χώρα σε αυτόν τον ορισμό. Αλλά από τον ορισμό που βλέπω είναι σαφές ότι είμαστε για εμείς φορολογικός παράδεισος. Ε, όμως πρέπει να είμαστε να υπάρχει διαφάνεια ω προ αυτό. Ε, με προβληματίζουν κάποιε τροπολογίε που έχουν ε, καταθέσει συνάδελφοι για τη διαγραφή για παράδειγμα, της ανάκλησης της τραπεζικής άδεια σε περίπτωση ε, φοροδιαφυγής, φορολογικής απάτης, κάτι το οποίο με εκπλήσει. Το ίδιο ισχύει ε, σε ό,τι αφορά την ε, τραπεζική μυστικότητα που υπάρχει, το απόρριτο, το τραπεζικό που υπάρχει στην Ελβετία, υπάρχουν προτάσεις να διαγραφεί, το οποίο μάλλον με προβληματίζει και διαγραφεί των ε, διατάξεων ε, υποβολής εκθέσεων αναχώρα. Ε, ελπίζω πραγματικά να μην υπερψηφιστούν τέτοιες τροπολογίες και να μείνουμε στις συμβαστικές που έχουμε συμφωνήσει. Έχω ένα ερώτημα προς την Επιτροπή, εφόσον παρευρίσκεται εδώ έτσι κι Ξέρουμε ότι εφόσον συζητούμε την ώρα που φυγεί και το καθεξής, υπάρχουν δύο σαφείς οδηγίες που έχουν δημιουργήσει προβλήματα και ήδη η Επιτροπή έχει επισημάνει ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει αναθεώρηση ε, και σε ό,τι αφορά αυτές τις δύο οδηγίες λοιπόν έχετε προχωρήσει στην... καθόλου στην αναθεώρησή τους και πότε πρέπει να περιμένουμε ε, την αναθεώρησή τους. Τέλος, ε, περιμένω τις τελικές διαπραγματεύσεις και είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Εντάξει. Θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή μετά τους ομιλητές, να έχουν και λίγο χρόνο στη διάθεσή τους να σκεφτούν. Κύριο Στρατσέκ, το ECR. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Τι Ωραία και σαρκαστική έναρξη της συζήτησης. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερως ε, μια τέτοια αρχή και αναμφίβολα το επιχείρημά σας ε, το εκφράσατε σε ένα φιλικό πνεύμα και έτσι δεν θα απαντήσω. Ίσως να σας εκπλήξω μάλιστα με κάποιες από τις δικές μου παρατηρήσεις σήμερα, αλλά όχι και πολύ, δυστυχώς. Κυρία εισηγήτρια. Προετοιμάσατε μια έκθεση που ε, αριθμεί την ε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους. Και έτσι, σε αυτή τη δομή θα βασιστώ και εγώ για να παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις. Που μου οδήγησαν να υποβάλω τις δικές μου τροπολογίες. Πρώτον, για την ε, φοροδιαφυγή περίπου 1-3 ευρώ ε, χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό είναι λυπηρό. Λυπηρό, κυρία Εκχάρτ. Είναι μια λέξη, ένας όρος που ίσως να σας εκπλήσει, εκ στόματός μου, και μέτρα μπορούν να ληφθούν ε, τα οποία εμείς τα επικροτούμε, τα χαιρετίζουμε τέτοια μέτρα. Χαίρομαι την παρατήρηση της κυρίας Γκουλάρ, η οποία δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, που τονίζει την αναγκαιότητα αποφυγής ε, απώλειας ε, εσόδων που προκύπτουν από την φοροδιαφυγή, ούτως ώστε τέτοια έσοδα να ε, οδηγήσουν στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Πολύ σωστή παρατήρηση, κατά τη γνώμη μου, την οποία μπορούμε να στηρίξουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εν γέννη συμφωνώ, ακόμα και με την κυρία Συγήτρια, που λέει ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να ε, ε, υποσκάψει την εμπιστοσύνη των ε, φορολογουμένων και των πολιτών σε ό,τι φορά την συλλογή φόρων. Αυτό είναι το σωστό. Σε ό,τι φορά την φοροαποφυγή τώρα, αυτό το σημείο μπορούμε να το εξετάσουμε από δύο οπτικές γωνίες. Πρώτον, ως άμεση συνέπεια της έλλειψης διαφάνειας δυσνόητων φορολογικών κωδίκων και της ε, υπερφόρτωσης ε, υπερβολικών ε, φοροαπαλλαγών και έτσι δίνουμε χώρο και έδαφος για την ανάπτυξη της φοροαποφυγής. Και δεύτερον, οι φορολογούμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις χειρίζονται το φορολογικό σύστημα και τα έσοδα από την φορολογία. Εγώ στις δικές μου τροπολογίες ε, αναφέρομαι στην ε, επιθετική φοροαποφυγή που είναι ανεπιθύμητη και δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Κάτι το ενδιαφέρον κατά την εξέταση των τροπολογιών ήταν ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ε, οδήγησε στην εκκίνηση ενός μεγάλου διαλόγου σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, κατά τη γνώμη μου, κάθε διαγωνισμό. Ε, κάθε είδους ανταγωνισμού είναι υγιής, ακόμα και σε ό,τι φορά τη φορολογία. Αυτά σε ό,τι αφορά την αντίθεσή μου προς ε, την εναρμόνιση του φορολογικού συστήματος. Τώρα, για τους φορολογικούς παραδείσους. Παρότι εγώ έχω καταθέσει τροπολογία που υπογραμμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ενεργά να ε, διαδραματίσει ρόλο σε επίπεδο G8 και G20 για την ε, διακυβέρνηση, για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συζητηθεί και να ε, συμφωνηθεί σε τέτοιο επίπεδο στο προσοχές μέλλον. Δεύτερον, για τον ε, νέο ορισμό του φορολογικού παραδείσου θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, σεβαστούμε τον ορισμό του ΟΣΑ, γιατί αποτελεί έναν κατάλογο κριτηρίων που, με τον οποίο συμφωνούν όλοι. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα δικό μας ευρωπαϊκό ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με τα χαράς ε, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση πάντα με μια φιλική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάντελ για την ΚΟΥ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μετά από την πρώτη συζήτηση που είχαμε δώσει στην Επιτροπή μας υπήρξαν καλές προτάσεις από την εισηγήτρια και έχει πάρει μια θετική τροπή η εξέταση αυτής της έκθεσης. Πολλά από αυτά που βρίσκονται στην έκθεση και στις συμβαστικές ε, τροπολογίες μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Θα ήθελα να πω όμως με σαφήνεια ότι όπως ελέγχθη από τους πράσινους, εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις διαγραφές οι οποίες έχουν γίνει στην έκθεση αυτή. Δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Εδώ θα πρέπει σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία της Επιτροπής μας θα πρέπει να πούμε ευθαρσώς ότι έχουμε σκεφτεί για το ποιε είναι οι καλύτερες προτάσεις για τα θέματα αυτά και πού πρέπει να αλλάξει η τωρινή κατάσταση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά δύο φορές στο παρελθόν. Όταν υπάρχει ένα δισεκατομμύριο ευρώ που χάνονται από φοροαποφυγή και φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή στην Ευρώπη, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι υπερβολικά απαλός. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια σε, βάθο, σε βάρος της κοινωνίας και γι' αυτό το λόγο οι πολιτικοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Μια δεύτερη παρατήρηση. Είναι καιρός ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε μια κρίση για να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ήδη και πριν από την κρίση ξέρουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τύχουν ρύθμιση και θα πρέπει να ελεγχθούν για να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στον χρηματοοικονομικό χώρο που αφαιρεί πόρους από την πραγματική οικονομία και την ε, <clears throat> κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν οι πλούσιοι να υπομισθούν ένα μεγαλύτερο βάρος από ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και όχι όλα αυτά να αναφέρονται στους φτωχούς. Αναφέρθηκε το θέμα του ανταγωνισμού, ότι είναι θετικό, αλλά αυτό δεν ισχύει για το φορολογικό τομέα. Γιατί είδαμε σε τι οδηγεί αυτό ο φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Αυτό τελικά αποβαίνει σε βάρο όχι μόνο των απλών πολιτών, των αδυνάμων δηλαδή στην οικονομία, αλλά και σε βάρο των ε, υποδομών στα κράτη-μέλη και γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε στην έκθεση αυτή να είμαστε σαφείς ότι η κάθε χώρα, η κάθε, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή και θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει ότι δεν θα αφήνει να γίνεται η φοροαπαλλαγή, η φοροδιαφυγή και ε, φοροαποφυγή Εν κατακλείδη μπορώ να υποστηρίξω πολλά από τα στοιχεία της ε, έκθεσης και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω επεξεργασία. Τώρα, με τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει το θέμα των ε, <clears throat> φορολογικών παραδείσων, ο κατάλογος του όσα είναι καλωσμένο, αλλά και εκεί θα πρέπει να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις, κατά την άποψή μου. Καλώς. Ο κύριος ε, Τερών έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω φιλανδικά. Είναι πολύ θετική η τοποθέτησή μας όσον αφορά την έκθεση. Είναι σημαντική. Η φοροαποφυγή και η φοροαπάτη είναι πολύ αρνητικά πράγματα. Ο φόρος είναι η βάση της πολιτισμένης κοινωνίας. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ποιος είναι ο στόχος της ε, έκθεσης. και τι πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα της φοροποφυγής και της φοροαπάτης. Θέλω να αναφερθώ στις αρχές που συμπεριλαμβάνονται στις δικές μου τροπολογίες που ελπίζω θα συμπεριληφθούν στις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν είναι προσπάθεια εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων αυτή. Όχι, θέλουμε να, επα... Ε, αυτό είναι θέμα επικορικότητας. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τη φορολογική πολιτική. Δεν θέλουμε να αυξηθεί ο δημόσιος τομέας και ας αυξηθεί το φορολογικό εισόδημα. Είναι καλύτερο να μειωθούν ε, τα ποσοστά της φορολόγησης. Πρέπει να επιτρέπεται και στο μέλλον η δυνατότητα ε, ανταγωνισμού μεταξύ των φορολογικών συστημάτων. Η φοραπάτη είναι το ερώτημα. Αλλά δεν θέλουμε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα χωρίς όμως να αλλάξουμε ριζικά τα φορολογικά συστήματα των χωρών. Ευχαριστώ η κυρία Λούλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ υπέβαλα κάποιες τροπολογίες. Δεν ξέρω όμως αν έχουν ε, γίνει αποδεκτές στις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες δεν έχω στη διάθεσή μου πρέπει να πω ότι δεν είχαμε το χρόνο να συζητήσουμε για το θέμα στην ομάδα μου. Δεν συζητήσαμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Υπέβαλα λοιπόν κάποιες τροπολογίες. Και αυτό διότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Σημερίζομαι, όπως και όλος ο κόσμος, την ιδέα ότι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει φόρους. Φόρους που προβλέπει η νομοθεσία να καταβληθούν. Και έχω πλήρη επίγνωση το ότι η χρηματοπιστωτική κρίση από την οποία περνάμε και δεν μειώνεται καθιστά ακόμα πιο αφόρητο το φαινόμενο της φορολογικής απάτης. Από αυτά που άκουσα μέχρι τώρα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφωνία επί των στόχων. Η συζήτηση αφορά περισσότερο τον τρόπο επίτευξης των στόχων. Για να προχωρήσουμε πιστεύω ότι όλοι θα ωφεληθούμε αν βασιστούμε επί αποδεδειγμένων, γεγονότων, περιστατικών, χωρίς να παίζουμε με νούμερα, με πολλά μηδενικά. Και να βασιστούμε περισσότερο στην εμπειρία. Καλύτερο αυτό παρά να κυκλοφορούν συνθήματα. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να συμφιλιώσουμε την προστασία του ιδιωτικού τομέα, της ιδιωτικής σφαίρας, με την πληρωμή των φόρων. Είναι απλούστατη αυτή η μέθοδος. Το σύστημα της φορολόγησης στην πηγή είναι κάτι απλό και αποτελεσματικό. Παραδέχομαι ότι η οδηγία για την φορολόγηση των καταθέσεων χρήζει βελτίωσης. Κι αν η φορολογική βάση είναι ευρύτερη, δεν θα είναι πλέον δυνατόν να ξεφύγει κανείς από το φόρο κάτι που συμβαίνει σήμερα. Να λέμε όμως ότι το τραπεζικό απόρριτο και η πληρωμή των φόρων είναι αντίθετα πράγματα νομίζω ότι δεν είναι ακριβές. Διαπιστώνω ταυτόχρονα ότι η Γερμανία που προασπίζεται την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Μιλώ εδώ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Εφαρμόζει το σύστημα της κράτησης στην πηγή των φόρων. Διότι αυτό το σύστημα είναι απλό. Ότι είναι απλό και αποτελεσματικό. Ε, νομίζω ότι είναι παράξενο αυτό ότι ενώ διαθέτουμε αυτή την ενιαία αγορά να συνεπάρχουν δύο διαφορετικά καθεστώτα ένα για τους Γερμανούς εντός της χώρας και άλλο σύστημα για τους Γερμανούς εκτός, στο εξωτερικό. Αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί ε, μια προφανέστατη αντίφαση και θα έλεγα ότι πρόκειται και περί ε, και κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πρέπει να υπογραμμιστεί είναι της αποδοχής της φορολόγησης. Μπορούμε να... Μπορεί να μας λυπείτε, όχι, αλλά είναι γεγονός ότι από ένα όριο και πέρα, ψυχολογικό όριο φορολόγησης, οι πολίτες δεν συμφωνούν πλέον. Και ε, από τη στιγμή που αισθάνονται ότι τους κλέβουν, ε, έχουν την τάση να κάνουν κολπάκια, να πηγαίνουν αλλού και να πηγαίνουν πιο καθαρότερους ουρανούς φορολογικούς. Και βλέπουμε, γίνεται μια παθιασμένη συζήτηση πάνω σε αυτό στη Γαλλία. Και αυτό το πρόβλημα δεν φωτίζεται επαρκώς, διότι ένας πολίτης πρέπει να δίνει στη χώρα 75, 80 των κερδών του με την πρόσθεση των διαφόρων φόρων δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού θα πρέπει οι πολιτικοί να το λάβουν αυτό υπόψη και να μην γίνεται κυνήγι μαγισσών που δεν οδηγεί παρά σε, στον φτωχαίνει η χώρα τους. Ε, τελευταία παρατήρηση. Νομίζω ότι για να είναι χρήσιμη αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να βασιστεί επί πληροφοριών επαληθευμένων, εξακριβωμένων, αδιαμφισβητήτων θα ήθελα να ζητήσω από την ε, εισηγήτρια να μην χρησιμοποιεί πολύ εύκολα συνθήματα, διότι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε και θα πρέπει να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε χωρίς να αναθεματίζουμε ένα τον άλλον. Και νομίζω ότι έχουμε χρόνο για να δούμε και τις συμβαστικές τροπολογίες. Πολλοί συνάδελφοι της ομάδας μου βλέπω ότι έχουν υποβάλει τροπολογίες. Και αφού συζητήσουμε, θα μπορούσα να σας πω κατά πόσο μπορώ να δεχτώ κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες ή όχι. Να ζητήσουμε από την Κομισιόν τα φώτα της <clears throat> και να απαντήσουν τα ερωτήματα. Ο κ. Ζούνεντοφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και την εισηγήτρια για το έργο που έχει φέρει σε πέραση υποστηρίζοντας το σχέδιο δράσης της Κομισιόν και τις συστάσεις τις οποίες διατυπώσαμε το Δεκέμβριο. Είναι κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα η υποστήριξή σας για να μπορέσω να σταθώ στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τον κύριο Έικοτ για το χρονοδιάγραμμα καταρχήν. Το χρονοδιάγραμμα για την ε, αναθεώρηση των οδηγιών που εμπλέκονται. Είναι μία από 34 δράσεις που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που ερεκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου και προβλέπεται να λάβει χώρα το 2013 αυτή η αναθεώρηση. Η ελπίδα μας είναι να μπορέσει να περατωθεί η διαδικασία αυτή μέχρι το φθινόπωρο. Και φυσικά ο αντικειμενικός μας στόχος είναι πέρα από τη γενική αυτή επισκόπηση σε, <clears throat> στα θέματα αυτά, θέλουμε να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο οι τωρινές οδηγίες είναι ε, λυσιτελείς για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ε, αναθεώρησης που θα φέρουμε σε πέρα σε φέτος και επιπλέον σε σχέση υπάρχουν, ε, οι, υπάρχουν ε, τα θέματα των ε, ανισομεριών, των υβριδικών ανισομεριών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα θέματα αυτά και επομένως όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην συνολική επισκόπηση που θα κάνουμε και ελπίζουμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα μπορούμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτή την αναθεώρηση και εφόσον μου έχετε δώσει το λόγο θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να τονίσω ότι εξετάσουμε με μεγάλη προσεκτική, πολύ, προσεκτικό τρόπο το θέμα των φορολογικών παραδείσων στην ε, σύσταση που διατυπώσαμε το Δεκέμβριο υπό την έποψη του ορισμού του τι είναι φορολογικός παράδεισος πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια στην περίπτωση αυτή που να μην είναι μόνο τα κριτήρια του ΟΣΑ αλλά και τα κριτήρια που εφαρμόσουμε εμείς στα δικά μας κρατη μέσα στον κώδικα συμπεριφοράς για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και επίσης εξετάζουμε προσεκτικά τα δυνητικά μέτρα στα οποία θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν με τα πρότυπα καλής διακυβέρνησης που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα να ισχύουν και της αντιμετώπισης παραβατικών ε, φαινομένων, να προτείνουμε μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν από τα κράτη-μέλη για να αλλάξουν συμπεριφορά. Επομένως, θα εξετάσουμε και πάλι αυτά που έχουμε προτείνει στην ε, σύσταση αυτή του Δεκεμβρίου. Παραμένουμε πιστοί σε αυτή την οδηγή γραμμή, οδηγό γραμμή και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και την ε, κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στι συστάσει τη Κομισιόν ήταν και σκόπιμα και σύμμορφα με τις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε απόψεις με το Κοινοβούλιο και να σας εξηγήσουμε περισσότερο την ε, επιχειρηματολογία μας και τον λόγο για τον οποίο έχουμε προτείνει όλα αυτά τα μέτρα και το γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε όλα τα μέτρα τα οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέταση και έχουν αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της ε, επεξεργασίας της προηγούμενης σύστασης. Δεν τα δεχτήκαμε τότε, αλλά μπορούμε και τώρα να επανέλθουμε και να εξηγήσουμε τις επιλογές στις οποίες προβήκαμε και γιατί ορισμένα στοιχεία δεν περιλήφθηκαν στο σχέδιο δράσης και στις συστάσεις μας. Δεν θα ανασταθώ εδώ μόνο. Um, Mr. that, that um, response... Κύριε Χαρτ, ικανοποιήστε τι ε, απαντήσει αυτέ εντάξει. Ας δώσουμε το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια ε, για να μας κάνει μια γενική επισκόπηση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αναφορά που έγινε για το 1-3 ε, ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο λόγω της ε, διαφυγής φοροφυγής και των φορολογικών παραδείσων προέκυψε από μια μελέτη ε, που κάλεσε ο κύριος Βέρφη. Ε, αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούν ακόμα και οι ίδιοι επίτροποι, επομένω. Ε, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο βέβαια να κάνουμε εκτιμήσεις και υπολογισμού, σχεδόν ανέφικτο. Όμως ε, είναι μια μελέτη που αναγνωρίστηκε από οικονομικούς ε, οργανισμούς και γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς, ε, αποφασίσαμε και μετά τη συνάντηση των σχεδόν να, να μείνουμε στους βασικούς ορισμούς της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού Ξέρω ότι υπήρχε συζήτηση για την φοροαποφυγή, αλλά η πλειοψηφία αποφάσισε να ακολουθήσουμε αυτόν τον ορισμό. Όμως μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, αν θέλετε, στο δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για τις συμβιβαστικέ. Όπως είπα και σήμερα το πρωί, υπόσχομαι να, να στείλω ε, τον δεύτερο γύρο συμβιβαστικών μέχρι αύριο το απόγευμα συμφωνώ με κάποιες από τις ε, προτάσεις σας, αλλά όχι με όλες, για να είμαι κι εγώ σαφής. Για τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων και τον ορισμό του ΩΣΑ. Συμφωνώ πολύ με τον ορισμό του ΩΣΑ, όμως αυτός ο κατάλογος είναι κενός αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο σε έκθεση της Επιτροπής Οίκων σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να πάει παραπέρα για να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνεισφορά ε, στον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Και απολογούμε απέναντι στους ε, σκιώδεις, γιατί στη συνάντηση μας δεν είχαμε χρόνο ε, να τα συζητήσουμε αυτά, τους ορισμούς και τις κυρώσεις για όσους μπαίνουν στο μαύρο κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Όμως αυτά τα δύο στοιχεία ε, πράγματι ταυτίζονται και μετά όσα αναφέρονται και στις, ε, στις συμβαστικές. Για την ανάκληση της, της ε, τραπεζικής άδειας, εδώ θα επιμείνω. Υπήρξαν κάποιες τροπολογίες, αλλά πραγματικά ήταν πολύ λίγες. Να διαγραφεί δηλαδή αυτή η αναφορά. Έτυχε μεγάλη στήριξη η πρότασή μου σε αυτό το θέμα. Βεβαίω και η φορολόγηση είναι θέμα που επίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά με τα τόσα χρήματα που χάνονται κάθε χρόνο και εγώ προσπάθησα να πάω λίγο παραπέρα. Και σε μια έκθεση υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ίσως να πρέπει να διαπραγματευτούμε λίγο με την Επιτροπή, σίγουρα με το Συμβούλιο Τουλάχιστον όμως έχουμε μια ε, καλή έκθεση, ένα καλό ορισμό και ένα ισχυρό μήνυμα εκ μέρους ε, της Επιτροπής Οίκων και του Κοινοβουλίου. Τότε μπορούμε να κάνουμε και αυτό το βήμα. Αλλιώς ε, έχουμε μια έκθεση άνευ περιεχομένου. Γι' αυτό θα επιμείνω στη σημασία αυτών των θεμάτων. και είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε και σε συμφωνία γιατί ήδη συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις και τις τροπολογίες που έχουν ε, καταβληθεί. Και χαίρομαι γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει στήριξη για να έχουμε μια ισχυρή έκθεση στο τέλος. Και προς την κυρία Λούλινγκ, δεσμεύομαι να, να σας στείλω απόψε ή αύριο το πρωί τον δεύτερο γύρο. Ε, αυτά. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και τους Χιώδης. Να υπενθυμίσω μόνο του συναδέλφους ότι 24 Απριλίου ψηφίζουμε και θα πάει στην Ολομέλεια τον Μάιο του 2013 βεβαίως. Εντάξει. Time. Προχωράμε πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο πρόγραμμά μας. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο. Έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 10 παρα 5 και βλέπω απουσία σκιωδών. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι πεντάλεπτο, αλλά μην το σκάσετε και αν βγείτε έξω να επιστρέψετε. Σας παρακαλώ.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

Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Προσπαθώ να μην χάνουμε χρόνο γιατί μερικές φορές τελειώνουμε νωρίτερα, μερικές φορές λίγο αργότερα και μας ξεφεύγουν κάποια θέματα, οπότε αν μπορούμε να συντονιστούμε το χρονοδιάγραμμα. Um, Είναι η δική μου έκθεση και προεδρεύω. Θα παίξω διπλό ρόλο. Θα προσπαθήσω. Ελπίζω να είχατε τη δυνατότητα να ρίξετε μια ματιά στην έκθεσή μου. Νομίζω ότι στην αρχική μου παρουσίαση προσπάθησα να σας δείξω την προσέγγιση που ήθελα να ακολουθήσω και τις αρχές που ήθελα να εφαρμόσω όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, έχω περιορισμένες δυνατότητες, δεν μπορώ να γράψω το αριθμό προτάσεων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν τώρα δυνατότητα οι σκιώδεις και τα μέλη της Επιτροπής να εκφράσουν ιδέες και προτάσεις. Ήθελα να σας πω ότι ήταν πολύ καλή συνάντηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ την περασμένη εβδομάδα. Θέλει πράγματι να υποβάλει σχετικές προτάσεις τον Ιούλιο και επιθυμεί να ξέρει ποιες είναι οι απόψει μας, ούτω ώστε να τις λάβει υπόψη, την άποψη και της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου. Άρα θέλω μια ευρεία συζήτηση. Ξεκινώντας, ακροθυγώς να συνοψίσω. Ποια είναι η προσέγγιση μου, θέλω να σας πω. Θέλω να δώσω χρόνο στους σκιώδεις να συζητήσουν και να παρέμβουν. Είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να την ακούσουμε. Όπως γνωρίζετε, Πέρσι, Φεβρουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων, ούτω ώστε να εξετάσει αν χρειάζονται πρόσθετε μεταρρυθμίσει των δομών του τραπεζικού σύστηματος τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα μειωνόταν η πιθανότητα έτσι να χρεοκοπήσουν τράπεζε και τον αντίκτυπο που θα είχε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνεχιστεί η ζωτική λειτουργία και αν χρεοκοπήσουν τράπεζες για να προστατευθούν οι πελάτες του λιανικού τομέα. Ε, καλωσόρισα λοιπόν την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου. Θεώρησαν και εκείνοι όπως και εμείς ότι υπήρχε υπερβολική ανάληψη κινδύνου, πολύ ψηλό επίπεδο μόχλευσης, πολύ μεγάλες απαιτήσεις εφαρμογή το κεφάλαιο και τη ρευστότητα, πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα το τραπεζικό και ήταν στη ρίζα της χρηματοστατικής ε, κρίσεως όπως γνωρίζουμε. Και πράγματι όμως πολλές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν. Η ομάδα όμως κατέληξε συμπεράσμα ότι οι περαιτέρω δομικές διαθετικές αλλαγές ήταν απαραίτητες και υπέβαλαν πρόταση ότι θα έπρεπε να υπάρξει νομικός διαχωρισμός κάποιων επικινδύνων χρηματοστατικών δραστηριοτήτων από, τις διάφορες, από διάφορα ταμιευτέρια που είναι στους ομίλους τους τραπεζικούς. Λοιπόν, ο διαχωρισμός ε, θέλει να καταστρήσει πιο ασφαλείς κάποιους κοινωνικά ευαίσθητους τομείς ε, και να περιοριστεί και η ε, διάσωση τραπεζών μέσω των χρημάτων του φορολογωμένου όπως και των καταθέσεων και χρήσεως των καταθέσεων διάσωση όπως βλέπουμε στην Κύπρο. Ο διαχωρισμός αυτός θα πλουστεύσει και θα κάνει διαφανέστερους τραπεζικούς μηχανισμούς και θα είναι πιο εύκολη η επίλυση προβλημάτων και η διάσωση και η εποπτεία. Θα πρέπει λοιπόν ο τραπεζικός τομέας να είναι πιο ανθεκτικός ε, αντιμετωπίζοντας χρηματοστικές κρίσεις. Θα πρέπει να μειωθεί το κόστος και ο κίνδυνος ε, από πλευρά των των τραπεζών όσον αφορά τα δημοσιονομικά και θα πρέπει ε, να είναι ασφαλές το περιβάλλον, να είναι αποτελεσματικό, να εξυπηρετεί τις ανάγκες πραγματικής οικονομίας, τους πελάτες, τους καταναλωτές και να στηρίζει την παροχή πιστώσεων στην οικονομία, κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις διότι εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε τον τομέα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για να αναπτυχθεί και η οικονομία. Τι έκανα λοιπόν, όπως είπα αρχικά. Ήθελα να βάλω κάποιες βασικές αρχές, να μειωθεί ο περίπλοκος χαρακτήρας του συστήματος, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να περιοριστεί η διασύνδεση μεταξύ των πιο επικινδύνων εμπορικών ε, δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων, να βελτιωθεί ε, η διαχείριση των διαφόρων επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε ένα υπεύθυνο σύστημα αμοιβών, διότι το σύστημα των αμοιβών και των μισθών του τραπεζικού συστήματος ε, ενθάρρυνε την ανάληψη πολύ μεγάλων κινδύνων. Θέλουμε αποτελεσματική ανάκαψη των τραπεζών, ενίσχυση του κεφαλαίου των τραπεζών, και να χορηγούνται πιστό στην πραγματική οικονομία. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη στοιχεία. Όχι μόνο για μια μεταρρύθμιση, αλλά για μια αλλαγή τη όλη νοοτροπία στο τραπεζικό σύστημα. Και πολλοί λένε ότι η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει. Και αν αλλάξει η κουλτούρα και η νοοτροπία, προφανώ εμπλέκεται και η αλλαγή των δομών. Συνεπάγεται και η αλλαγή των δομών. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. αν δείτε βαθμολόγηση των αγορών καταναλωτών που παρήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πίνακα το Δεκέμβριο του 2012 δημοσιεύτηκε. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο που υπήρξε ποτέ και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου. Να, τη θεωρήσουμε, να θεωρήσουμε αυτή την έκθεση σαν βάση της μεταρρύθμισης. Τώρα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που έχω στην έκθεσή μου που αφορούν τη δομή του πεζικού συστήματο. Και ελπίζω να σχολιάσετε, συνάδελφοι, να υποβάλλετε τροπολογίε, να προτείνετε βελτιώσει. Λοιπόν, ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή σε ένα σημείο. Και στην έκθεση Λικάνα αναφέρθηκε, αλλά και στη δική μου. Ποια είναι η βάση μα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ συγκεντρωμένο το τραπεζικό μα σύστημα. 14 όμιλοι ευρωπαϊκοί. Είναι πολύ ε, σημαντική συστημικά 15 ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν 43% των αγορών σαν αφορά τα στοιχεία ενεργητικού. 150% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσης αντιπροσωπεύουν και κάποια κράτη-μέλη ε, αναφέρουν και υψηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, το ποσοστό μεγέθους τράπεζα με ΑΕΠ έχει τριπεσιαστεί από το 2000 μέχρι τώρα και σε ενδιαφέρει τώρα στην κρίση την κυπριακή ότι τα στοιχεία ενεργητικού που υπολογίστηκαν από το ΔΝΤ το 2011 ήταν 835% του ΑΕΠ της ε, Κύπρου. Ε, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να καταρρεύσει, για να αποτύχει. Too big to fail. Ε, λοιπόν, χρειάζεται μια μεταρρύθμιση σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό συνεχώς βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των καταθετών ε, μετά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις ίσως καταλήξουμε σε μια κατάσταση που ανέφερε και ένα σχολιαστής. Δηλαδή, οι καταναλωτέ πρέπει να εμπιστεύονται την τράπεζα όπω εμπιστεύονται το γιατρό του. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα υγεία, υγείας, ε, όπω λέμε του τραπεζικού συστήματο. Μπορεί να εμπιστευτεί κάποιου γιατρού, έτσι. Ε, και πρέπει σε κάποιο βαθμό να πούμε ότι βλέπουμε περισσότερε αποτυχίε από ό,τι επιδόσει στον τραπεζικό τομέα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ανέφερα κάποιες αρχές για τη διεθνωτική ε, μεταρρύθμιση που χρειάζεται. Αν δείτε τα στοιχεία της μεταρρύθμισης, βασικό στοιχείο συζήτησης και θα εστιαστούν συνάδελφοι από αυτού, είναι ο διαχωρισμός. Πώς διαχωρίζουμε ε, νομικά πρόσωπα, δεν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε διαχωρισμό, διαχωρισμό σαν αυτό σκοπό, αλλά έχουμε κάποιο στόχο μέσω του διαχωρισμού. Στόχος, να μην υπάρχει διακοπή των δραστηριοτήτων τραπεζών και γιατί έχουμε κλείσιμο, κατάρρευση, κλείσαν οι τράπεζε μέχρι την Πέμπτη στην Κύπρο. Διότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να διαχωριστούν ε, οι επενδυτικέ δραστηριότητε από τι δραστηριότητε του Ελληνικού εμπορίου. Ένα από του στόχου ποιο είναι, να εξακολουθούν οι συναλλαγέ ακόμα ε, και αν υπάρχει μια κρίση στο σύστημα. Αν δείτε ε, τα επίκαιρα ζητήματα, αυτά που συμβαίνουν τώρα, Βλέπετε ότι δεν μπορούν οι διευθύντες σπιτιών να πουλήσουν την περιουσία τους στην Κύπρο. Έχετε τα ATM που δεν έχουν ρευστό να δώσουν, τράπεζες που έχουν κλείσει γιατί δεν θέλουμε να γίνουν μαζικές αποσύσεις από τις τράπεζες. Ε, αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα μη ε, βιώσιμου ανθυγινού τραπεζικού συστήματος ε, που οδηγεί προς την χρεοκοπία, οδηγείται προς την χρεοκοπία. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε κυρίως για τους καταθέτες. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέσω μεταρρυθμίσεως. Γι' αυτό χρειάζεται νομικό διαχωρισμός. Το πρώτο είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Θα έχουμε διαχωρισμέ πηγές χρηματοδότησης για το ελληνικό ε, ε, τομέα σε σχέση με τον επενδυτικό. Θα έχουμε όρια όσον αφορά το βαθμό που βασίζονται διάφοροι φορεί για χρηματοδότηση και δεν θα πρέπει να υπάρχει νομική βάση για μετακίνηση κεφαλαίου και ρευστότητα μεταξύ ομίλων κυρίως για να χρηματοδοτήσουν πιο επικίνδυνες δραστηριότητες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την πρόταση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σαφή κριτήρια που θα επιβάλλονται για το διαχωρισμό ε, και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το συστημικό κίνδυνο που δημιουργείται και για τους φορείς του λιανικού εμπορίου και για τους επενδυτικούς και για το τραπεζικό σύστημα γενικά για να έχουμε κάποια περιθώρια ασφαλείας, buffers για το κεφάλαιο. Λοιπόν, τώρα να πάμε στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που αναφέρθηκαν στην έκθεση της ομάδας ηλιοπιπέδου. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη μηχανισμή ελέγχου και διακυβέρνηση, καλύτερα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, να δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα. Θα πρέπει να υπάρχει αποκάλυψη των κινδύνων ε, και ιδέωσες κυρώσεις. Ε, το 2011, σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, Είχαμε περάσει ένα ψήφισμα για την ε, διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ζήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ψήφισμα της Ευρω... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 11η Μαου του 2011 και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει αυτό ότι θα οδηγήσει ανεξάρτητε αποφάσει ο διαχωρισμό και διακυβέρνηση για κάθε φορέα, διαφορετικά διαχωρισμό των διοικητικών συμβουλίων και των μελών των δύο φορέων και ξεχωριστού μηχανισμού υποβολή αναφορών και εκθέσεων. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στο συστήματα αμοιβών μισθοδοσίας. Θα θέλουμε να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί, ούτως ώστε οι αμοιβέ και η νοοτροπία αμοιβών ε, στις τράπεζες να δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, στη χορήγηση κινήτρων ε, με μεγαλύτερες περιόδους αν, αναβολών κυρίως για το μεταβλητό κομμάτι του μισθού ακόμα και μέχρι την εποχή συνταξιοδότηση. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα αμοιβών μισθοδότηση να δώσουν προτεραιότητα σε άλλα εργαλεία πέρα από την καταβολή ρευστού, παραδείγματο χάρη μετοχέ, συμμετοχή. Ε, θέλουμε τα συστήματα αμοιβών και μισθοδοσίας να αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις, να εστιάζονται επί της εξυπηρετήσεως των πελατών και μακροπρόθεσμη χρηματοστητικής σταθερότητα και όχι επί α, βραχυπροθέσμων κερδών. Βλέποντα τι κυρώσει θα πρέπει να ζητήσουμε αποτελεσματικέ κυρώσει που θα είναι αποτραπτικές και για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα και είπα ότι η δημοσίευση των επιπέδων των κυρώσεων και η ενημέρωση για τις κυρώσεις είναι ζωτική σημασία σαν αποτρεπτικό στοιχείο για εκείνους που παραβιάζουν τους κανόνες και βεβαίως ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει οι εποπτικές αρχές να έχουν την εξουσία αν είναι αναγκαίο και αντιμετωπίζεται κρίση οι εποπτικές αρχές εθνικές να μπορούν να εφαρμόσουν πλήρη νομικό διαχωρισμό των τραπεζών στο σύνολό τους. Όχι εντός του ιδίου τραπεζικού ομίλου. Αυτό θα βοηθούσε την ε, ανάκαμψη και την εκαθάριση. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω, που, διότι δεν είναι υγιές να έχουμε τράπεζες συγκεκριμένη χώρα που να αποτελούν το 835% το ΕΠ της χώρας. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό του τραπεζικού τομέα. Αν θέλουμε να έχουμε εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, θα πρέπει να προσφέρουμε διαφορετικές ε, τραπεζικές υπηρεσίες Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη ποικιλομορφία του τραπεζικού τομέα, να ενθαρρύνουμε μεγα... οι τράπεζες κινούνται προς τους ε, ε, καταναλωτές, να υπάρχουν διάφορα είδη ε, ε, τραπεζών και να υπάρχει δανειοδότηση μεταξύ ομοτήμων peer-to-peer -peer lending, όπως αποκαλείται, νέος τρόπος δανειοδότησης, κυρίως προς μικρές επιχειρήσεις, και θα ήθελα να δούμε πώς μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό και πώς μπορούμε να κινηθούμε προς αδειοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων, διότι όπως ε, είπα είναι πολύ καλές εναλλακτικέ ε, για μικρές επιχειρήσεις για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση. Και γι' αυτό ζήτησα από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι δικέ του εποπτικέ αρχέ να έχουν σαφή στόχο να προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στο τραπεζικό τομέα. Και ένα άλλο θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για του καταναλωτέ και το έθεσαν να το εξετάσουμε. Η διευκόλυνση τη αλλαγή τραπεζών για τον καταναλωτή θα είναι καλύτερο έτσι ο ανταγωνισμό αν οι καταναλωτέ αισθάνονται ότι μπορούν να μετακινήσουν του λογαριασμού του εύκολα για να έχουν καλύτερε συμφωνίε και καλύτερες ε, υπηρεσίες στον τομέα της λιανικής να μπορούν να το κάνουν. Άρα να μειωθούν οι φραγμοί ε, για να μπουν καινούργιοι ε, πελάτες σε τράπεζες και επίσης να αρθούν και οι φραγμοί για να αλλάξει ο άνθρωπος τράπεζα, να φύγει από την τράπεζα και να πάει σε άλλη τράπεζα. Λοιπόν, πάρα πολλοί τομεί χρειάζονται επεξεργασία, μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτούς, είναι σημαντικό και το συζήτησα με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ποιο θέλουμε να λειτουργεί η εσωτερική αγορά, υπάρχουν διασυνοριακές δραστηριότητε και στα 27 κράτη-μέλη, στον τραπεζικό τομέα, όμως πρέπει να σεβόμαστε και ότι έχουμε πολύ διαφορετικό, ποικιλόμορφο τραπεζικό τομέα. Πρέπει να σεβαστούμε την ποικιλομορφία και τη διαφορά. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύουν όταν αυτό ενδείκνυται το δικό του τραπεζικό του σύστημα. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ τα σχόλιά μου και θέλω να ακούσω κάποια σχόλια των σκιωδών και άλλων συναδέλφων της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Um, Η κυρία Λούλιν, κυρία Πρόεδρε. Έχω δει πολλά έγγραφα σε διάφορες ε, εκφράσεις, <clears throat> σε διάφορες γλώσσες, αλλά το έγγραφό σας υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς και να κάνει μια γενική συζήτηση. Είδα ότι υπάρχει στα γερμανικά, αγγλικά. Εγώ θα ήθελα να έχω κάποιες εξηγήσεις γιατί μπαίνει στη διάταξη μια έκθεση εάν είναι διαθέσιμη μονάχα στην αγγλική γλώσσα. Κυρία Λούλινγκ, λέει η πρόεδρο. Έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση και ίσως αμπουσιάζεται. Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια συζήτηση επί τη βάση του κειμένου στην αρχική γλώσσα, μια αρχική συζήτηση. Στη συνέχεια θα είχαμε της, ε, τη δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών σε διάφορες γλώσσες. Γι' αυτό τα έγγραφα που βλέπετε έχουν τροπολογίες σε ανάμεικτε γλώσσες. Αυτό είναι το θέμα του Γραφείου Καταθέσεων Τροπολογιών όμω, όχι δικό μας. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αποφασίσανε ότι για την αρχική τουλάχιστον συζήτηση θα παραμείνουμε επί τη βάση μονάχα του αγγλικού κειμένου. Δεν σημαίνει αυτό ότι αποκλείονται περαιτέρω συζητήσεις όταν τα κείμενα διαθέσιμα σε όλε τι γλώσσε. Δεν θέλω να καταργήσω τα δημοκρατικά σας δικαιώματα, κυρία Λούλινγκ, σίγουρα θα έχετε τη δυνατότητα να συμβάλλετε σε αυτή τη συζήτηση. Ζητώ απλώ την υπομονή σας, γιατί η Κομισιόν θέλει να καταλήξει σε μια πρόταση τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. μα ζήτησε να κάνουμε μια συζήτηση και να προχωρήσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Δεν θέλω να σας περιορίσω λοιπόν, αλλά θα πρέπει να δεχτείτε και σε αυτή τη διαδικασία. Κύριο Γκοζές. Δεν αναφέρουμε σε εσά ω εισηγήτρια, αλλά ω προεδρεύουσα στην Επιτροπή μα. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που λέει η κυρία Λούλινγκ. Το σύστημα αυτό με των γλωσσών γίνεται ένα οδοστρωτήρα που επιβάλλει παντού τα αγγλικά και εμποδίζει τη δημοκρατική συζήτηση. Μα ενδιαφερόμαστε για του πολίτε. Λέμε πρέπει να καταλαβαίνουν οι πολίτε. Αν πάνε στι ιστοσελίδε μα δεν έχουν καμία γλωσσική μορφή. Έτσι θέλουμε να φτιάξουμε την Ευρώπη. Μα είναι πολλοί που λένε είναι πιο οικονομικό να δουλεύουμε σε μια γλώσσα, να έχουμε τα κείμενα σε μια γλώσσα. Όχι, δεν είναι πιο εύκολο. Υπάρχει μια πολυμορφία. Αυτό θέλω να τονίσω. Μάλιστα, λέει η πρόεδρο. Θα καταγράψω τα σχόλιά σα. Και θα τα μεταφέρω στην ε, πρόεδρο και τη γραμματεία για να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι όλε οι γλωσσικές μορφέ του κειμένου θα είναι διαθέσιμε στο τέλο τη εβδομάδα. Κάνουμε την αρχική συζήτηση με την έκθεση με τη μορφή που έχει τώρα. Δεν πιστεύω ότι αυτό εμποδίζει το μέλη της Επιτροπής μας να ε, εκφράσουν την απόψή τους. Νομίζω ότι και έξω από την έκθεσή μου έχετε ήδη απόψη για τα θέματα αυτά και θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις ακόμα και αν δεν είναι συγκεκριμένες τροπολογίες στη δική μου έκθεση. Ξεκινώ λοιπόν και καταγράφω την αντίρρηση της, ε, τα σχόλια της κυρίας Λούλιν και του κύριου Κοζές. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου. Κυρία Βόρτμαν Κόλ και εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε ο Ζωάν Πολ και η Άστριντ για τις γλωσσικές μορφές των κειμένων. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με ταχαία βήματα για αυτή την έκθεση. Είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε την Κομισιό να προχωρήσει στην ε, πρόταση νομοθεσίας. Αλλά τούτου λεχθέντο θα πρέπει να ζητήσουμε και από τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου να επιταχύνουν το έργο του, ώστε να έχουμε όλε αυτέ τι εκθέσει στι μητρικέ μα γλώσσε. Γιατί αυτό είναι μια σημαντική συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να επιμείνω στο να περάσετε το μήνυμα προ την Πρόεδρό μα. Μπαίνω τώρα στο... <clears throat> στα θέματα ουσίας. Για μένα ένα κέριο θέμα που αναφέρεται στην εκθεσή σας είναι το κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός ορισμένων δραστηριοτήτων των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθεσία. Βλέποντας τις μεταρρυθμίσεις που είναι υπό εξέλιξη, νομίζω ότι ήδη έχουμε εγκρίνει την ε, οδηγία CRD4, την MIFID, την EMIR σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να, εξασ... να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση ΛΙΚΑΝΕΝ και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σαφή άποψη σε σχέση με τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται πέραν της νομοθεσίας που έχει ήδη εγκριθεί από μας. Είναι σημαντικό να το πράξουμε αυτό και επίσης είναι σημαντικό να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση ενός νομικού πλαισίου που θα προσδώσει ασφάλεια δικαίου σε όλους τους εμπλεκομένους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διερευνήσουμε περισσότερο σε αυτή την έκθεση. Πρέπει να έχουμε και κατευθυντήριες γραμμές που θα δώσουμε στις εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για να εξασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή του νομικού αυτού πλαισίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το τόνισα και την προηγούμενη φορά είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόσουν τη δική τους προσέγγιση επί τη βάση της δικιάς τους τραπεζικής δομής. Οι Γάλλοι έχουν μια άλλη αντιμετώπιση, οι Γερμανοί μια τρίτη, οι κάτω χώρες θα προτείνουν και αυτή μια διαφορετική δομή. Όλα αυτά μπορεί να βολεύουν σε εθνικό επίπεδο, να ταιριάζουν με τα εθνικά τους τραπεζικά συστήματα, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ τις ε, θηγατρικές και τα υποκαταστήματα των μεγάλων τραπεζών σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι μια ενιαία αγορά και για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Αν δεν μπούμε λοιπόν σε αυτό το επόμενο βήμα για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα δώσει σαφήνεια στον τραπεζικό τομέα, ο κίνδυνο είναι ότι θα παραμείνουμε σε αυτόν τον κατακαιρματισμό τη εσωτερική αγορά στα τραπεζικά θέματα και όχι να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη διαμεθοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Και αυτό μπορεί να είναι ακόμα και κάποιο κίνητρο για ορισμένα κράτη-μέλη να αποσυρθούν από ορισμένε δραστηριότητε αντί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μια ενιαία αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τι μεγάλε τράπεζε που είναι πιο πολύπλοκε, που έχουν πιο ευρείε δραστηριότητε συναλλαγών <clears throat> σε αξιόγραφα κτλ. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια σωστή ανάλυση αυτών των θεμάτων στην έκθεση Λικάνεν. Πιστεύω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βασιστούμε σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Η <clears throat> κατεύθυνση που παίρνει η έκθεση Λικάνεν είναι ότι τα σχέδια επίλυσης για τις τράπεζες, οι διαθήκες εν ζωή όπως λέγονται, πρέπει να είναι το σημείο κίνησης και πρέπει να είναι και το σημείο εκκίνησης όταν απαιτείται μια διαρθωτική μεταρρύθμιση αυτών των ε, τραπεζών και γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την προσέγγιση του κ. Λικάνε και της Επιτροπής του. Αν μπούμε τώρα όμως στη συζήτηση τι πρέπει να περιέχει αυτή η νομοθεσία και το νομοθετικό πλαίσιο. Όταν πρόκειται για το εμπόριο, για τις συναλλαγές που κάνει μια τράπεζα για δικό της λογαριασμό, το λεγόμενο proprietary trading, είναι κάτι το οποίο είναι σαφές, ότι πρέπει να διαχωρίζεται από την φυσιολογική τραπεζική διαδικασία. Αλλά όταν το δούμε αυτό σε θέμα ε, αριθμητικό, οι μεγάλες εταιρείες είναι τμήμα των, ε, του λιανικού τραπεζικού, των λιανικών τραπεζικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή είναι τμήμα της επενδυτικής, των επενδυτικών τραπεζών, των δραστηριοτήτων επενδυτικής τράπεζας. Πώς θα διαχωρίσουμε λοιπόν όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείε. Γιατί έχουν πολλές φορές οι μεγάλες εταιρείε που δεν είναι τράπεζες, έχουν δραστηριότητες που αφορούν αντιστάθμιση κινδύνου, ανταλλαγές ε, σε επίπεδο συναλλάγματο κτλ. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εξετάσει και ποιο είναι ο αντίκτυπο των αποφάσεων που θα πάρει. Και μετά, βλέποντα το περιεχόμενο τη έκθεσή σα, όταν δείτε την παράγραφο 9, παραδείγματο χάρη, ακολουθείτε την προσέγγιση ότι από τα αριθμητικά στοιχεία καθορίζεται τι είναι η λιανικού χαρακτήρα τραπεζική δραστηριότητα και ξεχωρίζεται αυτό το τμήμα των δραστηριοτήτων ή λέτε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε και την πολυμορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τις μεγάλες, ε, μεγάλες εταιρείες και κατά πόσο θα πρέπει μια τράπεζα να μπορεί να δίδει πλήρες υπηρεσίες στους μεγάλους αυτούς ε, επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα σε σχέση με την εκθεσή σας. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο τόνισα προηγουμένω, θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και της ε, εποπτικής αρχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λέτε εσείς ότι πρέπει να υπάρξει μια σαφής, ένας σαφής νομικός διαχωρισμός των δύο ειδών δραστηριοτήτων, αλλά προϋποθέτεται ότι αυτό είναι εύκολο να γίνει τη στιγμή που είναι πολύμορφος και πολυπίκυλο ο τραπεζικός τομέας. Εγώ θα σκεφτόμουν να υπάρχει ένας ε, διαφορετικός τρόπος προσέγγισης όπου οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα παίρνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, υπάρχουν φαιές περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να δώσουμε μία σειρά αρχών ως κατευθυντήρες γραμμές στους εθνικούς επόπτες και τους ευρωπαϊκούς επόπτες για να κάνουν σωστά τις ε, ενέργειες διαχωρισμού. Δεν πρέπει να με παρεξηγήσετε. Εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι ε, επικίνδυνου χαρακτήρα ενέργειες συναλλαγών όταν δεν έχουν χαρακτήρα αντιστάθμισης κινδύνου να περισταλούν. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα ερωτήματα να τα αντιμετωπίσουμε γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να εξυπηρετήσει την πραγματική οικονομία, κάτι το οποίο περιέχεται στους στόχους που θέλουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να επιτύχουμε. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Κάποια ακόμα σχόλια σε σχέση με το θέμα της εταιρική διακυβέρνησης. Και μάλλον πρωτού φτάσω εκεί, σε σχέση με το θέμα της ε, ε, εταιρικής διακυβέρνησης, είπατε ότι θέλετε να εφαρμόσετε τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Αλλά δεν το λέτε αυτό για την ε, διαρθρωμένη μεταρρύθμιση. Αυτό είναι θεληματικό να κάνετε διαφορετική προσέγγιση στους δύο αυτούς τομείς. Θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Και εξακολουθώ να έχω κάποια ερωτήματα με την προσέγγιση που προκρίνει η Επιτροπή Λί και θα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα για το κομμάτι της εταιρική διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε συμπληρωματικά μέτρα πέραν της το, τωρινής νομοθεσίας, δηλαδή του, της οδηγίας CRD. Τα θέματα της αμοιβή των στελεχών. Ποιος είναι ο στόχος σας για τα σημεία αυτά. Όταν λέτε ότι έχουμε εγκρίνει πρόσφατα ή θα εγκρίνουμε σήμερα την τελική συμφωνία θα έχουμε για την ε, οδηγία CRD. Και επίσης <clears throat> για τα θέματα της ε, διακυβέρνησης. Μιλάτε για τους εθνικούς ε, επόπτες εδώ αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρεται ο Εθνικός Επόπτης, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να αγωνιστούμε στο βαθμό του δυνατού να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, το Συμβούλιο πηγαίνει σε χίλιε άλλε κατευθύνσει. Αυτά είναι λοιπόν τα σχόλιά μου και προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση μαζί σα και με του άλλου συναδέλφου. Και είναι σημαντικό να παραμείνουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμα. δεν πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρήματα που θα την ε, βοηθήσουν να καθυστερήσει αυτήν την νομοθεσία. Για τα κράτη-μέλη ήδη προχωρούν και εμείς έχουμε χάσει χρόνο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προλάβουμε και να παίξουμε ηγετικό ρόλο με το να είμαστε γρήγοροι στην επεξεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Κλέντ από την Άλντα. Ευχαριστώ, Αλήν. Εμείς βλέπουμε πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεσή σου. Η διάγνωση, το γιατί καταλήξαμε σε μια κρίση είναι σωστή, αλλά είναι μόνο εν, μέρος, εν, μέρη ακρίβης, γιατί υπάρχουν και πολλά λάθη τα οποία έγιναν άμα σκεφτούμε την κρίση στην Ιλανδία, την κρίση στην Ισπανία, τις δυσκολίες της ε, Κύπρου. Αυτά δεν είναι θέματα υπερβολικής σημασίας της ε, επενδυτικής δραστηριότητας των τραπεζών υπήρξαν σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή το να υπάρχει διαχωρισμός της τραπεζικής δραστηριότητας από την επενδυτική δραστηριότητα δεν θα είχε οδηγήσει στο να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Επίσης, αναφέρεσε σωστά στο θέμα της ανάγκης να επανέλθει η εμπιστοσύνη που έχει χαθεί στο τραπεζικό σύστημα και να μην φορτώνεται πάντα ο φορολογούμενος με τη διάσωση των τραπεζών. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μία αντιμετώπιση η οποία δεν είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Έχουμε εισαγάγει πάρα πολλούς κανόνες, κανόνες ρευστότητος, κανόνες για την κεφαλουγική επάρκεια, κανόνες που απαγορεύουν τις ε, ακάλυπτες πωλήσει, όλα αυτά μπορεί να έχουν κάποια αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά. Αλλά θεωρούμε ότι έχει τελειώσει και περνάμε μέσα στο επόμενο επίπεδο, το να έχουμε εποπτικές αρχές κτλ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να κάνουμε μία ανάπαυλα και να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα και να έχουμε μία κριτική αξιολόγηση για το κατά πόσο ήταν θετικά και αποτελεσματικά όλα αυτά που έχουμε ήδη εγκρίνει και αν πρέπει να προσθέσουμε νέα στοιχεία σε αυτά, αν πρέπει να αλλάξουμε κάποια στοιχεία κτλ. Και έχουμε τώρα την ε, ε, έκθεση Λικάνεν, η οποία προέρχεται από ένα προβληματισμό που οδήγησε στον κανόνα Φόλκερ στις ΗΠΑ, αντίστοιχε ενέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Και εγώ νομίζω ότι είναι υπερβολικά έτσι, υπερβολική παρέμβαση αυτή η αντιμετώπιση που προτείνεται από την έκθεση Λικάνεν. Εγώ δεν ξέρω αν λύνει πραγματικά προβλήματα αυτή η προσέγγιση, γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι έχουμε μία λανθασμένη κουλτούρα διαχείρισης των τραπεζών, λανθασμένη κουλτούρα στελεχών των τραπεζών. Και αυτό αναφέρεις και εσύ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα και αυτό δεν είναι θέμα το οποίο θα μπορέσει να προκύψει από ένα νέο κανονισμό. Είναι μια μακρά διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Και πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να τροποποιήσουμε την προσέγγιση του κινδύνου στις τράπεζες, να έχουμε μια κουλτούρα υπευθυνότητο. Και μια διαρθωτική και μόνο ή φορμαλιστική αντιμετώπιση δεν γιατί για το ταπεζικό τομέα εγώ πραγματικά αμφιβάλλω αν θα βοηθήσει. Υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν γίνει και πάντα στον ακαδημαϊκό τομέα υπάρχουν όλο και περισσότεροι καθηγητές και ε, ειδικοί που διαλαμβάνουν τα θέματα αυτά λένε πολλές φορές ότι υπάρχουν, υπάρχουν ενδιαφέρουσες χάρη μελέτες που λένε ότι σε εμπειρικό επίπεδο έχει καταδειχθεί ότι στις ΗΠΑ η ύπαρξη ενός, ε, ενός μοντέλου παραδείγματος χάρη παγκόσμια τράπεζα, οικουμενικής τράπεζας που κάνει και επενδύσεις και λιανικέ δραστηριότητε, είναι κάτι το οποίο θα είχε βοηθήσει. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακριβή αυτή. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει μια λύση που είναι άσπρη ή μαύρη. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτά τα οποία γίνονται. Για μένα λοιπόν η πλήρης διαδικασία διαχωρισμού των τραπεζών σε επενδυτικό κομμάτι και σε κομμάτι λιανικής τραπεζικής δραστηριότητας είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό. Η έκθεση Λίκανε δεν αναφέρεται στην, στη δραστηριότητα επενδυτικής τράπεζας, αναφέρεται μονάχα στο εμπόριο το οποίο κάνει μια τράπεζα για δικό της λογαριασμό. Αυτό πρέπει να δια, διαχωριστεί από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Αλλά οι άλλες δραστηριότητες επενδυτικού χαρακτήρα δεν θέλει ο κύριος Λικάνεν να τις αποχωρήσει από την υπόλοιπη τραπεζική δραστηριότητα γιατί ξέρει ότι οι πελάτες χρειάζονται και αυτές τις υπηρεσίες. Ακόμα και οι μεσαίες εταιρείε είναι όλο και περισσότερο δραστηρίες ε, ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στι ΗΠΑ και αλλού. Και χρειάζονται λοιπόν όλε αυτέ τι τραπεζικέ υπηρεσίε από τι τράπεζε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιθανού κινδύνου κτλ. και να εξασφαλιστούν εναντί αυτών. Και επομένω κρατά μια κάπω πιο επιφυλακτική στάση επιπλέον. Όταν σκεφτόμαστε στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των τραπεζών, ερχόμαστε σε ένα θέμα που ο Γκούναρ Χέρκμαρκ είχε αντιμετωπίσει ως εισηγητής με την οδηγία αντιμετώπισης της κρίσης. Και προβλέπεται εκεί ότι όταν μια τράπεζα θεωρηθεί ότι δεν μπορεί πλέον να επιληθεί, πρέπει να υπάρξει εκεί ένας διαχωρισμός δραστηριοτήτων. Το αν πρέπει να το κάνουμε εκ των προτέρων αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να κάνουμε μια τόσο καθαρή διάκριση μεταξύ επενδυτική δραστηριότητα και κανονική τραπεζική δραστηριότητα. Παραδείγματο χάρη, πού θα βάλουμε τη διαχείριση κινδύνου στα θέματα αυτά. Πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο-τρει εβδομάδε, βγήκε μια δημοσίευση ε, από τον κύριο που καταλήγει ότι η λύση η λύση δεν είναι, να λέει ότι η λύση δεν είναι ο διαχωρισμός, αλλά απλώ οι τράπεζες να έχουν ε, επαρκές κεφάλαιο. Τη δεκαετία του 1910-1920 θεωρείται το δεδομένο ότι μια τράπεζα πρέπει να έχει ίδια κεφαλαία της τάξης του 20-25%. Και άμα σκεφτεί κανείς αυτά που κάνει η Ελβετία, η Ελβετία πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μεγάλες δύο ελβετικές τράπεζες τους έχει ζητηθεί να αυξήσουν πολύ περισσότερο το μετοχικό του κεφάλαιο και να έχουν περαιτέρω εργαλεία τα οποία λειτουργούν σε μια, κατα... σε μια κατάσταση κρίσης ως ίδιο κεφάλαιο και μπορούν να αυξήσουν το όριο του ιδίου κεφαλαίου στα 20%. Γι' αυτό σας λέω, εκφράζω και πάλι το σκεπτικισμό μου για τις ε, υποχρεωτικές προτάσεις υποχρεωτικού διαχωρισμού. Αν σκεφτείτε τώρα τις ε, μεγάλες γενικές τράπεζες, την Deutsche Bank, τη Societe Generale κτλ. Αν διαχωρίσουμε πλήρως και απόλυτα την δραστηριότητα επενδυτικής τράπεζας από τις τράπεζες αυτές, καταλήγουμε τελικά να έχουμε μία τράπεζα η οποία είναι σημαντική σε επίπεδο συστημικό, να έχουμε δύο τράπεζες που είναι σημαντικές, γιατί ακόμα και το επι το επενδυτικό κομμάτι μιας τέτοιας τράπεζας να πέσει σε δυσκολίες και αυτό θα έχει συστημική σημασία. Όσο δεν έχουμε λοιπόν ένα ταμείο επίλυσης ή ένα σύστημα ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις, απλώς πολλαπλασιάζουμε τους φορείς που μπορούν να βρεθούν σε δυσκολίες. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο με τον διαχωρισμό δημιουργούμε συνθήκε για να υπάρχουν τράπεζε που δεν θα μπορούμε με λογικό τρόπο να χρηματοδοτήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε την επίλυσή του. Ένα τελευταίο λοιπόν σχόλιο. Δεν πρέπει να πέσουμε λοιπόν στο σφάλμα να θεωρήσουμε ότι η διαδικασία λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών είναι αφεαυτής χωρίς κίνδυνο. Είδαμε τι έγινε στην Ισπανία. Με το να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό λοιπόν δεν ε, βγάζουμε από τη μέση τελείω τον, ε, τον κίνδυνο. Τέλος για τα κίνητρα. Είπα ορισμένα πράγματα για την ε, εταιρική διακυβέρνηση, αλλά για τα μακροχρόνια κίνητρα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί όπως έχουμε στην CRD4, ε, την οδηγία αυτή, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Έχουμε πει ότι πρέπει να περιορίσουμε τα πριμ, τα μπόνους των στελεχών που λέμε ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν το βασικό του μισθό το πολύ πολύ δύο φορές με την, με την θετική άποψη των μετόχων μιας ε, τράπεζας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός είναι ένας στόχος που μάλλον φαίνεται να μην επιτυγχάνουμε. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε η προλαλήσασα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την ε, αξία των εθνικών εποπτικών αρχών. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Αν είχαμε μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, σίγουρα δεν θα είχε φτάσει η κατάσταση στην Κύπρο στην κατάσταση που είναι σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια και αυτές οι αρχές να κάνουν σωστά την εργασία τους. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι το μαγικό ραβδάκι το να χωρίσουμε ε, απόλυτα τις ε, δραστηριότητες επενδυτικές από την κανονική τραπεζική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Um, Mr. Lamberts, the Greens. Ο κύριος Λάμπερτς από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Ελίν. Ναι, συνάδελφοι, θα συμφωνήσω με αρκετά τα όσα είπες, θα διαφωνήσω με κάποια άλλα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Λίκανεν ε, παρήγαγε εξαιρετικά ποιοτικό έργο, τόσο ενδιαφέρον μάλιστα, που εξετάζοντα και τη σύνθεση της ομάδας ε, είναι εξαιρετικά εξισορροπημένο ως έργο. Υπήρξε λοιπόν εκπροσώπηση από όλους ε, τους τομείς, από, από τον κλάδο, από τις εποπτικές αρχές, από τους καταναλωτές και έτσι είναι αρκετά εξισορροπημένη αυτή η έκθεση. Βλέπω γιατί λέτε ότι δεν πρέπει να προσθέσουμε το ένα ε, επίπεδο νομοθεσία μετά το άλλο χωρίς να σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο. Πράγματι ε, δικαιολογείται η ανάληψη δράσης σε αυτό το τομέα. Να σας δώσω το εξής επιχείρημα. Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια ανταγωνιστική ε, οικονομία της αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εφόσον έχουμε πλέον ιδρύματα που θεωρούν ότι, που αυτοποκαλούνται too big to fail, ότι είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν πλέον να καταρρεύσουν και με τέτοιους θεσμούς και φορείς πλέον δεν βρισκόμαστε στην οικονομία της αγοράς. Έχουμε ε, αν θέλετε, ε, που έχουν μια θέση στην αγορά που δεν δικαιολογείται απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Πριν μερικές ημέρες, ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, ένας ε, εκπρόσωπος του, Ευρωπαϊκού Ταμείου, του ευρωτανικού Ταπείου Οικονομικών ρώτησε τον κύριο Πρόκτο, συμφωνείτε Απαντήστε με ένα ναι ή ένα όχι. Συμφωνείτε ότι η τράπεζά σας θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τις ε, δραστηριότητες της στην αγορά χωρίς να χαίρει του πριμ ε, που οφείλεται σε έμεση δημόσια εγγύηση. Η απάντηση ήταν όχι, δεν θέλω η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες μας, θέλω μόνο μια επιδότηση μια στήριξη. Και αν δείτε και τις μελέτες που έχουν ε, διεξαγάγει ακαδημαϊκοί ε, στο, για το επίπεδο των, ε, της στήριξης που χαίρουν τέτοιοι οργανισμοί, βλέπουμε ότι το μέγεθος της δημόσιας επιδότησης ισοδυναμεί με τα κέρδη τους. Δηλαδή, αν δεν είχαν αυτή τις δημόσιες επιδοτήσεις, δεν θα είχαν κέρδη. Αυτό για μένα αποτελεί στρέβλωση της αγοράς. Και μια, ένας τέτοιος κλάδος ε, της οικονομίας που είναι τόσο θεμελιώδους σημασίας, νευραλγικός τομέας, θα πρέπει να λειτουργεί με όρους ε, ανταγωνισμού της αγοράς, όχι με επιδότηση τύπου Σοβιετική Ένωσης. Όχι, αλλά κοιτάξτε πώς ήταν το σύστημα ε, στη Σοβιετική Ένωση. Είχαμε την Κεντρική Τράπεζα που χορηγούσε τη ρευστότητα προς ε, τις ε, κρατικές τράπεζες που ε, λειτουργούσαν στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Αυτό βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο σήμερα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά η Κεντρική Τράπεζα δίνει ρευστότητα σε όλες τις τράπεζες της Ευρώπης που λειτουργούν όλοι και περισσότερο ως καρτέλ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι κατά την σύσταση του υποπτικού μηχανισμού και κατά την κατάρτιση των κριτηρίων που και εκεί για να διασφαλίσουμε ότι οι πιο σημαντικές τράπεζες θα υπόκειται σε επιτήρηση, σε, επί... σε επίπεδο ECB, Κεντρικής Τράπεζας, φτάνουμε στο 85% των ε, συνολικών ε, στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και από πλευρά οικονομία τη αγορά, λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση. Μάρτιν Έφελγη και Άτα Μάτια είναι ακαδημαϊκοί για τους οποίους ε, τρέφω μεγάλο σεβασμό και συμφωνώ ότι το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε ε, πολύ αυστηρούς κανόνες ε, μόχλευσης ρευστότητας και κεφαλαίου. Όμως, ε, Βίκη, δεν είναι αυτά που θέλαμε ακριβώς. Θέλαμε πιο αυστηρούς κανόνες και θέλαμε να θέσουμε υψηλά τον, τον πύχη. Θέλαμε λοιπόν ισχυρούς κανόνες σε ό,τι αφορά τη μόχλευση σε κάποια επιτύχαμε, σε κάποια όχι λοιπόν. Και σε έναν βαθμό επιλύουμε, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Αν ε, καταστούν αυτοί οι κανόνες ε, προοδευτικοί. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ε, συνάντησα κάποιους εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα της Γαλλίας και είπαν, ναι ξέρετε, εμείς πρέπει να ανταγωνιστούμε την JP Morgan, την Goldman Sachs, ε, την Morgan Stanley όπως και να έχει λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να μας αφήσετε να γίνουμε εξίσου ισχυροί με εκείνου. Δηλαδή να είμαστε υπεράνω κυβερνήσεων και δημοκρατίας. Αυτό μας ζητούν και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Για τις προτάσεις Λίκαναν, κατά πόσο είναι σωστές ή όχι. Ε, εφόσον ε, αφορούν τις, ε, τις, τα μεγάλα ιδρύματα, μπορεί να παραμείνει μια τράπεζα, αυτή η παγκόσμια οικουμενική τράπεζα, χωρίς να ξεπερνά όμως ένα μέγεθος. Αυτός είναι ο βασικός όρος. Και πάλι είναι θέμα μεγέθους. Αν μια τράπεζα γίνει υπερβολικά μεγάλη για να καταρρεύσει, αυτός για μας σημαίνει ότι είναι υπερβολικά επικίνδυνη για να υπάρξει και ασύμβατη με την οικονομία της αγοράς. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ε, παίρνω το μέρο των φιλελευθέρων ε, ω προ την αγορά και πρέπει να επιστρέψουμε στον ανταγωνισμό. Όχι, δεν αστείευομαι. Θέλω τον ανταγωνισμό γιατί ε, θα μας ε, οδηγήσει στην χρηστή συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την αγορά και πραγματική παραγωγή και δημιουργία αξίας. Όχι μια απλή άντληση επιτοκίων. Έτσι, οι τροπολογίε μου σε αυτό το ύφο θα κυμαίνονται. Μίλησα για την οικονομία της αγοράς, όμως ε, θα ήθελα να τονίσω και την ανάγκη της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη. Και εδώ έχω πραγματικές επιφυλάξεις, γιατί από την αρχή, έχουμε, από την αρχή της κρίσης έχουμε δει κατακαιρματισμό, αυξανόμενο κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς ε, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τι έγινε στην Κύπρο, το Σαββατοκύριακο. Ήταν ε, η πιο ανεύθυνη απόφαση που έχει λάβει ε, μια τέτοια ομάδα ε, λεγόμενων υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και ελπίζω θα του το πούμε και αυτοπροσώπους, αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο κατακρεματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που έχουν ως στόχο ιδρύματα που είναι κατά βάση διασυνοριακού χαρακτήρα. Ε, στη Γαλλία, σε πολλές χώρες. Τέτοια μέτρα θα κατακαιρματίσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την αγορά, ιδίως ε, για ιδρύματα που είναι διασυνοριακά, θα είναι πιο δύσκολο για μας ε, να ρυθμίσουμε τη δραστηριότητα αυτών των ιδρυμάτων. Γι' αυτό, Wolf, Ακόμα και μόνο για αυτό το λόγο πρέπει να πω ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δράση. Γιατί αν μείνουμε αδρανεί, ουσιαστικά λέμε στου Γάλλους, στους Γερμανούς ότι θέλουμε, ε, θέλατε να αποφύγετε την ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση και τα καταφέρατε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε κοινού κανόνε. Γιατί εδώ αντιμετωπίζουμε ιδρύματα ε, με πανευρωπαϊκή δράση και αντίκτυπο. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, όχι σε επίπεδο μεμονωμένου κράτου μέλου, ακόμα και αν πρόκειται για το μεγαλύτερο κράτο Αρκετά είπα σήμερα. Θα υποβάλω τροπολογίε ε, σε αυτό το πνεύμα. Προσβλέπω σε ενδιαφέρουσε συζητήσει. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά κοινά σημεία, αρκεί να συμφωνήσουμε ότι δεν θέλουμε δημόσια εχέγγυα για τις εμπορικές δραστηριότητες και ότι θέλουμε τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Um, I have uh, other speak- Λοιπόν, έχω και άλλους θέλω το λόγο. Λίν και άλλους. Sorry, well, Vicky, if you could just ask your group that whenever we, you change someone, we just need to know that, because I would have brought you in. Λοιπόν, αν ήξερα πιο νωρίς θέλετε να μιλήσετε, σας έδινα το λόγο, αν θέλετε να μιλήσετε για το ECR. Η Βίκη να μιλήσει πρώτα εκ μέρους της ομάδας. Δεν είχα υπόψη μου ότι άλλαξε σκιώδης για την ομάδα. Δεν αλλάξαμε το σκιώδη, αλλά έχω μια δήλωση εκ μέρου του Σαΐντ και ένα-δύο δικά μου σχόλια. Εκ μέρου του Σαΐντ. Λέει, είμαι πολύ ικανοποιημένο με την, το σχέδιο εκθέσεω. να είναι ξεκάθαρο ότι είναι απαραίτητο οι τράπεζε να ωφελούνται για επιδότηση άμεση ή έμεση του φορολογουμένου. Πολλέ προτάσεις συζητήθηκαν όπως η, οι οδηγία της κεφαλικής και άλλε αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Διαχωρισμό του τομέα λιανικού και χωδικού εμπορίου είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσω περαιτέρω στον Αμένο Βασίλειο. Ε, εισάγουμε σφυρίε απαιτήσει για προστασία και θέλουμε να εξετάσουμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό και ποια, ε, τι μπορεί να λύσει αυτό το θέμα του ring fencing, ring fencing της προστασίας. Λοιπόν, η ομολογία μας πρέπει να εξετάσει το θέμα πρέπει να εδράζεται η ενιαία αγορά επί ισχυρών θεμελίων χρηματοστατικών, θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει ούτω ώστε το βαθμό του δυνατό δεν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να σώσουν ε, ε, χρεοκοπούσε τράπεζε. ορίζει τι συστάσει τη ηγητρία για ε, αυξημένη εταιρική διακυβέρνηση. Θέλω να συζητήσω με άλλε ομάδε τη δυνατότητα να επανεισαχθούν τροπολογίε που θα εξετάζουν σε ποιο βαθμό οι διαδεθειά πρότυπα, τα EFRS, τα πρότυπα υπονομεύουν τη χρηματοστική σταθερότητα. Πολλοί επενδυτές ανησυχούν για το ρόλο που παίζουν τα πρότυπα για τα λογιστικά του ελλείμματος και η απομάκρυνση από την ορθή διαχείριση των τραπεζών ε, πώς οδηγεί σε χρηματοστοιχείες κρίσεις. Θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά για να κάνουμε συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σκιώδεις και οι συγητές και μαζί με όλη την Επιτροπή θα ήθελα να δω ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποφελές για τους πελάτες, είτε είναι άτομα, είτε είναι επιχειρήσεις, άρα χρειάζεται σωστή διαχείριση του κινδύνου, σωστά επίπεδα διαφάνειας και θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα κίνητρα. Να προσθέσω κάνα δύο δικά μου σχόλια. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην Κύπρο δείχνουν ότι και τα πλούστρα τραπεζικά μοντέλα μπορεί να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλους κινδύνους και όταν αντιμετωπι... κινδυνεύουν οι καταθέσεις υπάρχει μεγάλη κατακραυγή από το κοινό και μεγάλες πολιτικές πιέσεις για την προστασία των απλών καταθετών. Πέραν αυτού πρέπει να σταματήσει και η επιμόλυνση. Οπότε η πίεση επί των πολιτικών να παρεμβούν σε ένα απλό μοντέλο για τους καταθέτες είναι διαφορετικό από αυτό που αφορά άλλα κομμάτια τραπεζικού συστήματος. Κατά την άποψή μου ε, γίνεται σημαντικότερο το έργο που ο Χόκμαρ ε, κάνει όσον αφορά την ε, σαφήνεια των μέτρων και πώς μπορούν να συμμετέχουν οι μεγάλοι μέτοχοι στις όλες προσπάθειες. Απογοητεύομαι πολύ για τις διαπραγματεύσεις για το CRD, διότι η θέση αυτής της Επιτροπής όσον αφορά τη δυνατότητα να μπορούν να μπουν ε, διάφοροι μέτοχοι για να διασώσουν τράπεζα πριν μπουν δημόσια χρήματα, δεν συζητείται στον τριμερή διάλογο και για μένα αυτό ήταν από τα σημαντικότερα αιτήματά μας και καλύπτεται. Εξετάζεται μία ρήτρα η οποία είναι Τώρα, η σταδιακή εφάρμοση φορά την προστασία, το ring fencing. Καταλαβαίνω αυτό που αναφέρεται, ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει ποικιλομορφία τραπεζικό σύστημα και πρότεινα ότι ίσως δεν θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία λύση και μοναδική, αλλά είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεση μιας τράπεζας για να επιληθεί μία προστασία, ένα ring fence ίσως κατά τράπεζα να είναι κάτι που, να εφαρμόζεται κατά περίπτωση για τις αμοιβέ. Όλα όσα έγραψε Αιλίν ε, με βρίσκουν σύμφωνοι. Χρειάζονται μακροπρόθεσμα κίνητρα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ομόλογα και μετοχές και όχι ρευστό όσον αφορά να συνδέεται η μακροπρόθεσμη επίδοση με τη μακροπρόθεσμη αμοιβή επανειλημμένα. Είχα πει ότι μπόνους σε όριο ε, θα αυξήσει τους μισθούς σε ρευστό και αυτό άρχισε ήδη να συμβαίνει από τον τελευταίο τριμερή διάλογο για το CRD και όρια ανώτατο για τα μπόνους ίσως να κάνει βαρύ στις πληρωμές αντί ο πιστοβαρής ε, και αυτό είναι το προηγούμενο που ανέφερες. Δεν θέλει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο. Ε, η Ελίν. Α, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ρύθμιση των αμοιβών για τις τράπεζες δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς επακριβώς που δεν έχουν τους ίδιους κινδύνους, ε, που δημιουργούνται ηθικούς κινδύνους και που δεν συνεπάγονται και διάφορα πολιτικά προβλήματα που είναι παρόμοια με τον τραπεζών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Αλέν. Εγώ θέλω να επενέσω την ποιότητα και το ύφος της έκθεσής σου ή μάλλον της έκθεσης Αρλίν Μακάρτη. Έρχεται στην κατάλληλη στιγμή αυτή η έκθεση, σε μια χρονική στιγμή όταν πολλές χώρες έχουν κάνει αυτή την έκκληση για τραπεζική μεταρρύθμιση. Και θέλω να υποστηρίξω αυτά τα οποία ανέφερε η Κορίν Βόρτμαν Κόλ και ο Φιλιπ Λάμπερτς το γεγονός ότι πρέπει η προσέγγιση μας να είναι ευρωπαϊκή και αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους. Και για να βελτιώσει τα κείμενα που έχουν εγκριθεί στη Γαλλία και στη Γερμανία και τα οποία είναι υπερβολικά άτολμα σε σχέση με αυτό το οποίο είναι στις ΗΠΑ και σε σχέση με αυτά τα οποία προτείνει η έκθεση Λίκανεν. Πολλοί συνάδελφοι επανήλθαν στα διακυβευόμενα στο κείμενο αυτό, στα κείμενα αυτά. Από τη μία πλευρά θέλουμε να μειώσουμε την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες οι οποίες είναι too big to fail, υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν. Και ο Φίλιπ Λαμπέρς το τόνισε. Θα πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο την έμεση δημόσια εγγύηση των δραστηριοτήτων αυτών των ε, τραπεζών και δεύτερον θα πρέπει να κόψουμε τον, να μειώσουμε τουλάχιστον τον ομφάλιο λόρο που συνδέει την λιανική τραπεζική δραστηριότητα με άλλες δραστηριότητες που είναι λιγότερης ωφέλειας, ας το πω έτσι, για την οικονομία. Και επίσης πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα του ανταγωνισμού. Αλλά όχι να, αυξήσουμε τον ανταγωνισμό με το να μειώσουμε το μέγεθος των τραπεζών αλλά γιατί πρέπει να έχουμε και ενιαίου κανόνε ανταγωνισμού στι ευρωπαϊκέ χώρε. Γιατί αν κάποιε χώρε προβαίνουν σε τραπεζικέ μεταρρυθμίσει και κάποιε όλε, κάποιε όχι, δεν έχουμε ίσε συνθήκε ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο για να έχουμε πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι κατακαιρματισμός. Για τη μεταρρύθμιση στον τραπεζικό τομέα αυτό, αν δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν πολλές δυνατότητε. Υπάρχει αυτή, αυτό που κάνουν οι, οι Αμερικανοί με τον κανόνα Φόλκερ, δεν είναι, είναι φανερό. Δεν είναι αυτό που έχει στο κεφάλι του ο Επίτροπος Μπαρνιέ και δεν είναι αυτό το οποίο πρότεινε ο κύριος Λικάνεν και άλλοι στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο κανόνας Φόλκερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί καλύπτει κάποιες δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ ρισκαρισμένες, επικίνδυνες αλλά Όλα αυτά αφορούν και τη λεγόμενη σκιώδη τραπεζική ε, δραστηριότητα η οποία, της οποίας η ρύθμιση στην Ευρώπη είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα για μας η προσέγγιση του κυρίου Λικάνη. Συζητήσαμε μαζί του πριν από δύο εβδομάδες περίπου και συζητήσαμε λεπτομεριακά με αυτά μαζί του. Όταν βλέπει κανείς την έκθεσή του, έχει δύο προτάσεις. Αυτή που αναφέρει ο, ο Βολφ Κλίντ, ότι θα αυξήσουμε τις απαιτήσει για ίδιους πόρους των τραπεζών μέσα στο μοντέλο οικουμενικής τράπεζας και αν θέλουμε τώρα να κάνουμε δραστηριότητες οι οποίες είναι πιο ρισκαρισμένες θα πρέπει να αυξηθούν οι απαιτήσει σε ίδια κεφάλαια. Αλλά δεν αυτή που προτιμά ο κ. Λικάνεν. Αυτή που προτιμά ο κ. Λικάνεν είναι να ουσιαστικά να διαιρεθεί σε υποκαταστήματα μια μεγάλη τράπεζα, να χωριστούν οι δραστηριότητες να παραμείνει στο χώρο, της τραπεζικής επισκόπησης το, να περιληφθεί μάλλον στην τραπεζική επισκόπηση και ένα σύνολο από δραστηριότητε που βάσει του κανόνα Φόλκερ δεν θα, δεν θα βρισκόταν σε επισκόπηση. Αυτό το οποίο θέλει λοιπόν ο κ. Λίκανεν είναι να αντιμετωπιστούν πλήρως οι σχέσεις μεταξύ της Μητρικής Τράπεζας και του επενδυτικού βραχίωνα αυτής της ε, τράπεζας, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τον ομφάλιο λόρο. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση Μαρκάτη, γιατί κατά τη δική μου άποψη προχωρά ακόμα περισσότερο και από τον κύριο Λικάνεν. Αυτό το οποίο προτείνει είναι να υπάρξει αυτή η διάκριση σε διάφορα επίπεδα και να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων μεταξύ της μητρικής ε, τράπεζας και του επενδυτικού βραχίωνά της. Αυτό το βρισκό πολύ ενδιαφέρον. Όταν συζητάμε με τον κύριο Λικάνεν στις, στους διαδρόμους, το λέει αυτό, λέει ότι αυτό είναι μια ιδέα που δεν είναι στην εκθεσή του, αλλά λέει ότι είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία γύρω από την έκθεση Μακάρδιν, γιατί όπως ελέγχθη προηγουμένως, αν δεν γίνει τίποτα μέχρι τον Ιούλιο από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι φανερό ότι δεν θα έχουμε κανένα αντίκτυπο για όλα αυτά. Και για το θέμα αυτό το, της μετάφρασης των εκθέσεων, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αυτό. Εγώ ως γαλλόφωνος ενοχλούμε από την επικυριαρχία των Αγγλικών. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι πρέπει η Κομισιόν να προτείνει ένα κείμενο πριν από τον ε, Ιούνιο και αν δεν βιαστούμε δεν θα έχουμε τίποτα. Είναι πολύ απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν να μπορέσει να εκφέρει γνώμη και με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία για αυτή την νομοθεσία που σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο και έχει συμβολικό και εμβληματικό χαρακτήρα για τους συμπολίτες μας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πέτρε και κυρία Συγγήτρια βεβαίως, ακούσαμε όλους τους συναδέλφους ε, που μας ενθαρρύνουν να μιλήσουμε τη μετρική μας σήμερα. Αυτό θα κάνω και εγώ λοιπόν σήμερα. Στο τέλος όμως θα προσθέσω και μερικά σημεία στα αγγλικά. Να πω τα εξής. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε ένα θέμα. Δεν θα τεθεί λοιπόν τέλος στο μέγεθο τη νομοθεσία που μπορούμε να παράξουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται όχι, δεν υπάρχει. Τέλος. Είδαμε και τον κύριο Μπαρνιέ, έχει ε, περίπου 35 προτάσεις και αρκετέ προτάσει ε, από αυτέ που έχουν αναφερθεί και σήμερα ούτε καν έχουν καταρτιστεί ακόμα. Και όμως πριν καν ε, καταρτιστούν, πριν καν ε, τις διαβάσουμε και δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Και μάλιστα πολλές ε, ξεπερνούν τα επίπεδα G20. Μιλάμε για ακόμα ένα επίπεδο νομοθεσίας. Έτσι δεν είναι ο ρόλος μας εδώ στο Κοινοβούλιο να πούμε φτάνει μέχρι εδώ, να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της νομοθεσίας της εφιστάμενης. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Κάποιοι με επικρίνουν γιατί έχω πολύ φιλικές σχέσεις με τις τράπεζες, κάτι το οποίο δεν ισχύει, αλλά όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πράγματι πιστεύω ότι χρειαζόμαστε καλές τράπεζες. Δεν μπορεί να είναι όλες ε, κακές. Ευθύνη μας λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εξισορροπημένη ε, νομοθεσία, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ε, και για την προστασία των καταναλωτών, αλλά να έχουμε και μια αγορά που λειτουργεί σωστά. Ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Λίκαναν είπε, είπε ότι υπάρχει έδαφος περαιτέρω ανάλυσης ε, για τις επιπτώσεις των όσων προτείνονται εδώ. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι γενικά συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως και κλείνοντας ε, να πω ότι θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε ο Φίλιπ. Ο Κέινς δεν ήταν ε, που είπε ότι τελικά είμαστε όλοι φιλελεύθεροι ή όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη ρίση ε, για να βρούμε συνένεση με τους πρασίνους. Πραγματικά θα ήθελα να το ακούσω αυτό γιατί η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό. Και ο ανταγωνισμός χρειάζεται και στήριξη ισχυρών πολιτικών δυνάμεων όπως είναι η δική σου. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Φερέιρα. Well, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω αγγλικά. Όχι ότι διαφωνώ με την κυρία Λούλινγκ. Απλώς νομίζω ότι είναι πιο απλό σε περίπτωση τεχνικών συζητήσεων. Ξεκινώντας να πω ότι το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι ότι έχουμε πολλά επίπεδα νομοθεσίας. Και εδώ απαντώ αμέσως στον κύριο Σμιτ. Συμφωνώ ότι έχουμε πολλή νομοθεσία, όμως το θέμα δεν είναι να έχουμε το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε όλα και περισσότερη νομοθεσία. Είναι κατά πόσο ε, είναι απαραίτητη αυτή η νομοθεσία. Και δεύτερον, κατά πόσο είναι συνεκτική, συναφής. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για μένα. Για την νέα αυτή νομοθεσία θεωρώ ότι την χρειαζόμαστε σίγουρα. Και εδώ συμφωνώ με το λίμενο ότι ε, πρέπει να υπάρξουν σε ξεκάθαρες ενδείξεις. Δεύτερον, για τη συνοχή των όσων κάνουμε, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία. Ενώπιον και της Αιλίν. Έλεγα προηγουμένως ότι χρειάζεται αυτή η συνοχή Ποιο είναι το όραμά μας λοιπόν ε, κατά την εξέταση αυτού του ζητήματος. Στην εσωτερική αγορά ε, δεν θέλω να επαναληφθώ, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της έγκαιρης δράσης. Να μην ε, περάσει πολύ καιρό και οι Βρετανοί να υιοθετήσουν μια νομοθετική πράξη, οι Γάλλοι άλλοι, οι Σουηδοί άλλοι. Προφανώς όλοι αυτή η νομοθεσία είναι απαραίτητη γιατί τα κράτη-μέλη προβαίνουν στη θέσπιση τέτοιων νομοθετικών πράξεων. Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Αλλιώς ε, θα υπάρξει διαχωρισμός ε, στην ε, εσωτερική αγορά και δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός αν υπάρχει διαχωρισμός στην αγορά. Έτσι επιλύεται το ζήτημα της αναγκαιότητας για τη συνοχή πρέπει εδώ να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των στόχων μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την εικόνα, πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι για τα όρια της προσέγγισής μας ε, κατά την προσπάθειά μας να διασώσουμε και να εξηγειάνουμε ε, τις ε, τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως και τα όρια που έχουν αυτά τα, τα μέσα διάσωσης όταν προσπαθούμε να διασώσουμε μια τράπεζα που ουσιαστικά δραστηριοποιείται στον το, λιανικό τομέα. Υπάρχει λοιπόν όριο στην, ε, στις δυνατότητές μας σε ό,τι αφορά αυτές τις τράπεζες. Και προφανώς και αυτές τις τράπεζες μπορούν να έχουν προβλήματα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Όμως ε, τα εργαλεία στα οποία βασιζόμαστε έχουν ε, περιορισμένες δυνατότητες. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε συνοχή μεταξύ της ε, ε, προφύλαξης ε, των καταθέσεων και της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και από την άλλη πώς επιλύουμε το πρόβλημα των ρηψοκίνδυνων δραστηριοτήτων όπου είναι πιο αποτελεσματικές και οι προσεγγίσεις της διάσωσης. Πρέπει λοιπόν να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και πού ακριβώς θέλουμε να καταλήξουμε με ένα ε, σύστημα παρόμοιο του FDIC στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Δηλαδή όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα, οι καταθέσει και ε, η δραστηριότητα του τραπεζικού συστήματος ε, την εγγυήσεων. Όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει στη δική μα περίπτωση με τα μέσα που αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική σύνδεση με άλλα στοιχεία. Πρώτον, πώς, κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε στο καθεστώς ε, εγγύησης των καταθέσεων και ποια είναι η εξέλιξη ε, της νομοθεσίας ε, σε ό,τι το καθεστώς φύλαξη των καταθέσεων. Και το δεύτερο στοιχείο είναι οι εξελίξεις ό,τι αφορά την ε, ε, ενιαία εποπτική αρχή και την ενιαία αρχή, ενιαία αρχή εξυγίανσης. Συνοχή θα πρέπει να υπάρχει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέγεθος των τραπεζών. Συμφωνώ ότι μια χώρα δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για, τις, ε, για την τραπεζική δραστηριότητα που υπερβαίνει το μέγεθος του ΑΕΠ της κατά 8 φορές. Όμω ποιο θα είναι ο κανόνας ε, που θα εγκαθιδρύσουμε όταν δεν θα υπάρχει αρχή εξυγίανση και ε, αρχή εποπτείας που θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο ε, ή σε ευρωπαϊκό. Εκεί θα πρέπει να εξαλογίσουμε και πάλι την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού. Όταν θα πρέπει να περιορίσουμε το μέγεθος των τραπεζών βασίζεται σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με το μέγεθος της ε, χώρας ή το μέγεθος της τράπεζας συγκρίνεται με τη δυνατότητα του φορέα ε, εποπτείας και την ισχύ ε, του Ταμείου Εξυγένσης και της Αρχής Εξυγένσης. Γιατί ιδάλλως έχουμε εντελώς διαφορετικές τραπεζικές δομές, όχι βάσει ε, του μεγέθους της εσωτερικής αγοράς ή των κανόνων ανταγωνισμού, αλλά βάσει του μεγέθους των χωρών όπου έχουν την έδρα τους σε αυτές οι τράπεζες. Και αυτό μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτά ήταν μερικά στοιχεία που θα ήθελα εγώ ε, να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση γιατί η δική μου επιφύλαξη δεν είναι κατά πόσο αυτή, είναι αναγκαία αυτή η νομοθεσία, αλλά κατά πόσο συνάδει αυτή με την ευρύτερη δράση μας. Δύο παρατηρήσεις. Συμφωνώ απολύτως με την παράγραφο 15, όπου λέει ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την πρόσβαση των καταθετών ε, στους πόρους και να προστατεύσουμε ε, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πώς είμαστε τεθειμένοι να τα κάνουμε αυτό Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν, ε, ένα δίκτυο ασφαλείας. Και δεύτερον, για την παράγραφο 26 έχω μια συγκεκριμένη παρατήρηση. Πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να ε, προβλέψει διατάξεις ε, όχι μόνο για τους εθνικούς εποπτικούς φορείς, αλλά και για τους αρμόδιους φορείς. Γιατί εφόσον αναφέρουμε ότι θα έχουμε ενιαίο ε, εποπτικό φορέα, προφανώ αυτό θα είναι ο αρμόδιο και θα έχει μια τεράστια διαφορά στον ε, τρόπο προσέγγιση των τραπεζών. Και εκεί συμφωνώ με την ε, πρόταση τη συγγήτρια. Ευχαριστώ. Χόκμαρκ, uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση, διότι τονίζει κάποια από τα συζητούμενα. Εγώ είμαι διστακτικός, πώς να σας το πω όχι μόνο για αυτή την έκθεση, αλλά για αυτό που κάνουμε. Ίσως να ακούγεται ηρωνικό αυτό που λέγω. Τώρα προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα που ρυθμίζονται. Και αν κάτι κινείται στους στόχους μας και αυτό θα το ρυθμίσουμε. Ό,τι βλέπουμε να κινείται το ρυθμίζουμε. Και η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν είναι θέμα της οικονομίας αλλά της νομοθεσίας. Και κινούμεθα παράλληλα σε πολλαπλά μονοπάτια προσπαθούμε να λύσουμε ε, τα ίδια προβλήματα και δημιουργούνται προβλήματα συνοχής. Είναι σημαντικό βέβαια να θυμόμαστε ότι χρειάζεται μεγάλη χρηματοδότηση η ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε οι τράπεζες κάποια φορές να είναι απόλυτα ασφαλείς και καμιά φορά να αναλαμβάνουν δανειοδιωτώντας ε, κινδύνους. Από τη στιγμή που δανείζει κάποια χρήματα μια τράπεζα, αναλαμβάνει κάποιο κίνδυνο. Και όσο πιο νέα είναι η εταιρεία, μεγαλύτερο ο κίνδυνο. Μπορεί να είναι μικρή εταιρεία να έχει κίνδυνο, μεγάλη επιχείρηση που αναλαμβάνει κινδύνου, μεγάλου κινδύνου, μικρού κινδύνου, πάντα κινδύνου. Και θέλουμε να αναλαμβάνονται αυτοί οι κίνδυνοι. Και έτσι διαρωτώ με τι βγήκε από την ομάδα Λίκανεν. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ επένδυσεων και τομέα λιανικής δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είδα να υπάρχει ε, πρόβλημα ορισμού αυτού. Μιλάμε για το πρόβλημα της Κύπρου τώρα. Και σίγουρα δεν είναι η ανάμεξη μεταξύ επενδυτικών δραστηριοτήτων τραπεζών και λιανικού εμπορίου. Στην Κύπρο βλέπουμε να έχει τεράστια προβλήματα το μέσο της λιανικής στις τράπεζες. Πρέπει όμως το τομέα της λιανικής και καταθέσει καταθέσεις να χρησιμοποιούνται για κάτι. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο του μέλλοντος. Κάποιοι από εμά το πιστεύουμε. Εγώ όχι. Πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα δίνει σαφήνεια. Πλαίσιο για το αποδεκτό και το μη αποδεκτό. και έχουμε και το πρόβλημα των διαφόρων νομοθεσιών. Έχουμε το σύστημα εγγύσεως των καταθέσεων που εφαρμόζεται ε, και ελπίζουμε τελικά καταλήξει σε επιτυχή εφαρμογή. Και μετά έχουμε και το τέταρτο, τέταρτο οδηγία για τις κεφαλουχικές απαιτήσει ε, που ελπίζουμε να οδηγήσει σε ασφάλεια. Έχουμε την έκθεση της οποίας εισηγούμε εγώ για την ε, επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και πώς οι διάφορες αρχές εξετάζουν τις διάφορες τράπεζες και, βρίσκουν, και εξετάζουν κατά πόσο είναι φερέγγες. Άρα ε, ποια τράπεζα μπορεί να στηριχθεί και ποια δεν μπορεί να στηριχθεί. Ε, θεωρούμε ότι μέσω διαχωρισμού ε, τράπεζα που ασχολείται με το λιανικό τομέα από την τράπεζα που ασχολείται με τον εμπορικό τομέα ότι ο διαχωρισμός βοηθά την επίλυση των προβλημάτων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουν το εξή, ότι μπορούν να αναπτυχθούν, να ευημερούν οι τράπεζε, να πληρούν τι ε, νομικέ απαιτήσει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όχι να καθορίζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο. Το πρόβλημα της χρηματοδοτικής κρίσεως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι είχαμε επενδυτικές τράπεζες, ε, είχαμε ότι η ίδια τράπεζα ασχολιόταν με τις επενδύσεις και με τον τομέα της λιανικής, ότι αυτό οδήγησε στο πρόβλημα. αν κάποιες τράπεζες ε, μπορούν να ασχοληθούν μόνο με τη λιανική διατρέχει κάποιο κίνδυνο διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίσως το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο που θα οδηγούσε στην ευημερία τους. Ποιο είναι το πρόβλημα. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε νομοθεσία για, τις, ε, για την εγγύηση των καταθέσεων για, την, ε, για, την, ε, για τις κεφαλουχικές απαιτήσεις, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και την αναδιάρθρωση στη γενική του τραπεζικού τομέα πρέπει να το δούμε πιο ψύχρεμα. Να βάλουμε προτεραιότητες. Να έχουμε τους ακρογωνιαίους λίθους για την ενιαία αγορά πριν προχωρήσουμε πιο πέρα. Το πρόβλημα της τράπεζας δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί με το διαχωρισμό να επιληθεί. Και από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Από τη στιγμή που κανένα δεν μπορεί να μου αποδείξει ότι εδώ έγκυται το πρόβλημα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ε, προσέγγιση. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να πω αυτό. Κυρία Εισηγήτρια, συγγνώμη που διαφωνούμε ε, όσον αφορά την αφετηρία. Αυτό ήθελα να σα πω. Δεν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, λέει η Πρόεδρος. Ας προσπαθήσουμε να διεξέλθουμε αυτά τα ζητήματα. <clears throat> Αυτό το οποίο θέλω να κάνω <clears throat> είναι με τη βοήθεια της γραμματείας, επειδή δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα στη σύντομη αυτή έκθεση, ζητώ από τη γραμματεία να κάνει ένα σύντομο σημείο για το περιεχόμενο της έκθεσης Λίκανεν. Γιατί από κάποιες από τις απαντήσεις που άκουσα σήμερα, υπάρχει κάποια σύγχυση μάλλον στο μυαλό ορισμένων για το τι ακριβώς προτείνει η Επιτροπή Λίκανεν. Είναι μεγάλο το έγγραφο σε μήκο, είναι πολύπλοκο, πρέπει όμω να καταλάβουμε καλά τι λεπτομέρειε του τι περιέχεται. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω μεμονωμένα σε όλου του βουλευτέ, αλλά έχουν φύγει πολλοί και <clears throat> δεν έχει νόημα να κάνει κανεί ε, συζήτηση όταν λείπουν οι περισσότεροι. Ελπίζω ότι οι συνεργάτες σας θα μεταφέρουν αυτά που θα πω λοιπόν στους ε, βουλευτές που έδωσαν ερωτήματα ή έκαναν σχόλια. Εγώ νομίζω ότι με όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει είπε η κυρία Βορτμακόλ, νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε μονάχα μία εθελοντική προσέγγιση, πρέπει να έχουμε μία νομικά δεσμευτική δομή, γιατί σε μία εθελοντική δομή θα διαλέγει ο καθένα ό,τι θέλει και δεν θα έχουμε ενία αγορά. Θα γίνεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα. <clears throat> Επομένω, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο καθένα διαλέγει τι θέλει και δεν πρόκειται για το ότι ακολουθεί διαφορετική οδό το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, όπω είπε και η κυρία Βόρμαν Κόλ. Οι κάτω χώρε σκέφτονται αν θέλουν να κάνουν διαφορετικέ αλλαγέ τώρα. Και κάποιο το έχει αναφέρει αυτό στην τελευταία μα συζήτηση. <clears throat> Είχαμε <clears throat> ρύθμιση σε πολλού τομεί, κεφαλογική επάρκεια κτλ. Μήπως όμως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό να πούμε πριν από τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε πρώτα τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση και μετά αν είχαμε κάνει αυτό τα θέματα του κεφαλουχικής επάρκειας ή ρευστότητας θα είχαν ήδη ρυθμιστεί και δεν θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα στοιχεία νομοθεσίας. Λοιπόν, το γενικό θέμα της δομής του τραπεζικού τομέα ίσως θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα που θα αντιμετωπίζαμε και όλα τα άλλα τα επιμέρους θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν εκ των εστέρων. Ίσως κάποια από αυτά δεν θα χρειαζόταν να τα αντιμετωπίσουμε τόσο ενδελεχώς. Θέλω να με σαφείς επίσης για το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση πολλές φορές. Δεν μιλάμε για πλήρη, για πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων των κομματιών της τράπεζας. Μιλάμε για δραστηριότητες και δεν μιλάμε και για πλήρη διαχωρισμό δραστηριοτήτων στον τραπεζικό τομέα. Λέμε απλώς ότι πρέπει να γίνονται σε διαφορετικούς λογιστικούς λογαριασμούς, όπου επιβάλλονται οι κανόνες για τις τράπεζες. Είπε ο κ. Κλίντς ότι υπήρχαν αποτυχίες, αστοχίες τραπεζών που είχαν μονάχα λιανικέ δραστηριότητε και επομένω δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τον επενδυακό τομέα. Και λέει το πρόβλημα είναι η κουλτούρα των τραπεζών. Μα αυτό είναι και ένα λόγο για να έχετε μια ένα διαχωρισμό γιατί δεν πρέπει να αλλάξει κανείς, δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά με νομοθεσία. Η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει μονάχα με διαρθωτική μεταρρυθμίση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Αν δεν αλλάξετε την κουλτούρα αυτή, εκεί έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κλίντς, έχουμε προβλήματα στον τομέα λιανικών δραστηριοτήτων, αλλά γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχει διάκριση και η κουλτούρα του υπερβολικού κινδύνου, της ανάληψης υπερβολικού κινδύνου στον επενδυτικό τομέα, μεταφέρθηκε στις λιανικές ενέργειες. Γι' αυτό είχαμε λανθασμένες ενέργειες ε, προϊόντων λιανικής στους καταναλωτές, αλλά αυτό γιατί μπήκε το πνεύμα του κινδύνου από τον επενδυτικό τομέα μεταφέρθηκε από τους ανθρώπους αυτούς στον τομέα των λιανικών προϊόντων. Αν θέλετε λοιπόν να προ... προστατεύσετε, και εδώ πρέπει να ρωτήσουμε αν θέλουμε, τι θέλουμε να προστατεύσουμε, αν δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, θέλουμε να προστατεύσουμε τη δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στα λεφτά τους, να μπορούν ακόμα να δανείζονται από τις τράπεζες, να αγοράζουν και να πουλούν όταν θέλουν κάτι, τώρα έχουν παγώσει τα πάντα. Όλα έχουν σταματήσει γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες πολυπλοκότητες και ένα τέτοιο κουβάρι μεταξύ του επενδυτικού τομέα και του τομέα λιανικών δραστηριοτήτων που δεν μπορεί κανείς να τα ξεμπλέξει. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια μορφή διαχωρισμού, όχι τραπεζών, αλλά διακρίσεων. Δεν με πειράζει που η Deutsche Bank θέλει να είναι 75% επενδυτική τράπεζα και μόνο 25% να λειτουργεί στο λιανικό επίπεδο. Αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτό όμω δεν μπορούν να κάνουν. Είναι να έχουν τον κίνδυνο και στον επενδυτικό τομέα και στον τομέα λιανικού, λιανικών δραστηριοτήτων. Όσο κίνδυνο μπορούν να αναλάβουν, ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει το φορολογούμενο ή τις κυβερνήσεις που θα πρέπει να υπομισθούν τον κίνδυνο αυτό. Αν θέλω λοιπόν να παίξω στα χρηματιστήρια σαν επενδυτής, εντάξει. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσω ότι αν έχω υπερβολικούς κινδύνους, δεν πρόκειται μετά να πληρώσει την ύφη ο φορολογούμενος. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Φιλίπ, ότι υπάρχει μια υπόρρητη μορφή επιδότησης. Αν κανείς θέλει να υποστηρίξει την ενιαία αγορά, δεν μπορεί να θεωρεί αυτή η επίδοση η επιδότηση να δίνεται από τους φορολογούμενους. Αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τον κίνδυνο θα πρέπει να πληρώσει και την ύφη στο τέλος. Για μένα αυτό είναι απόλυτα λογικό. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτική, να μην πάρουμε αποφάσεις οι οποίες είναι ε, καθοριστικές, αλλά να διατηρήσουμε τη λειτουργία του συστήματος, αλλά να το κατευθύνουμε προς μια κατεύθυνση που να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και αν υπάρχουν κίνδυνοι από τον επενδυτικό βραχίωνα τη μια τράπεζα, αλλά αυτά να μην έχουν σαν αποτέλεσμα να καταραγώσουν και τον τομέα λιανικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Το άλλο σημείο είναι το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε την ενιαία αγορά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι κάποια κράτη-μέλη θέλουν να, προστατεύσουν το τραπεζικό του σύστημα και δεν θέλουν να καταλήξουν σε μια κατάσταση που εξακολουθούν να αναλαμβάνονται τεράστιοι κινδύνοι που τελικά καταλήγουν στα χέρια των φορολογουμένων και των κυβερνήσεων. Είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια δομή και ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι διατηρούμε και στα πλαίσια αυτής της προστασίας την ενιαία αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει ο στόχος αυτός που νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν αυτό Πρέπει να το σκεφτούν όλοι οι συνάδελφοι. Δεν το έχω αναπτύξει λογικά και σε μεγάλη έκταση. Είναι λογικό όμως ότι αν υπάρχει απώλεια στον ιδιωτικό τομέα, αυτές οι απώλειες πρέπει να καλύπτονται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει οι επενδυτές να βγάζουν κέρδη όταν τα πράγματα κάνει καλά και όταν τα πράγματα πάνε στραβά τότε πρέπει να είναι οι καταθέτες, οι φορολογούμενοι που επομίζονται τις ζημίες. Αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη αγορά θα πρέπει να δεχτούν ότι δεν έχει νόημα οι, οι τράπεζες να παίρνουν μονάχα την καλή μεριά και να αποκομίσουν τα κέρδη ενώ μετακυλίουν τις ζημίες τους ε, φορολογουμένους. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα, δεν έχω καιρό να αντιμετωπίσω όλα τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Θα ζητήσω από τη Γραμματεία να μας δώσει ένα υπόμνημα για το τι ακριβώς προτείνει η ομάδα Λικάνεν δεν προτείνει να αλλάξουμε τα πράγματα που κάνουν οι τράπεζές μας η ομάδα Λικάνη. Δεν θέλει να αλλάξουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αλλά λέει απλώς δεν μπορούμε να περιμένουμε ο φορολογούμενος να επιδοτεί τις τράπεζες. Αν παίρνουν υπερβολικό κίνδυνο οι τράπεζες δεν πρέπει να καταλύει στους φορολογούμενους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μορφή κινδύνου αναλαμβάνεται από τις τράπεζες, αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει την ασφάλεια των καταθέσεων. Δεν είναι αυτή η κατάσταση σήμερα στην, τράπεζα, στην Κύπρο. Δεν λειτουργούν οι τραπεζικές δραστηριότητες καθόλου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση κρίσης, εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα χρήματα για τους καταθέτες και τους φορολογούμενους. Και ότι μπορούν οι πολίτες να έχουν τις, τα λεφτά τους από την τράπεζα και τα λεφτά τους δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα Δομή και διαθέσεως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχω τώρα το χρόνο να σα πω πολλά περισσότερα. Ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε και μια πιο μακροσκελή συζήτηση, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει. Κύριε Χρόκμαρ, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, εγώ θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπατε, γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι κανένα από εμά θέλει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν για τι απόλυσεις του τραπεζικού τομέα. Ακριβώ αυτό θέλουμε να πετύχουμε με την νομοθεσία που θέλουμε να εφαρμόσουμε όχι μονάχα είχαμε τις κεφαλουχικές ε, ανάγκες, το CRD4, αλλά για τα θύματα ανάκτησης και επίλυσης σε περίπτωση αστοχίας μιας τράπεζας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι μέτοχοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρίσκο καταρχήν, μετά οι ομολογίουχοι, οι επενδυτές της τράπεζας. Αν θέλουμε τώρα αυτό να το χωρίσουμε σε κομμάτια, αυτό είναι πολύ παράξενο. Γιατί αν μια τράπεζα έχει σε ένα χώρο τις επενδυτικές δραστηριότητες και σε ένα άλλο χώρο της ε, λιανικού χαρακτήρα δραστηριότητες, ποιος θα αναλάβει τον κίνδυνο για την ε, επενδυτική δραστηριότητα για μένα, είναι η μέτοχοι. Σε μια μεγάλη τράπεζα είναι πιο πολλοί μέτοχοι. Αν έχει πολλές δραστηριότητες, έχετε πιο, πιο πολλούς ε, ε, μετόχους που μπορούν να απορροφήσουν τις απώλειες. Και υπάρχουν πιο πολλές επενδύσεις. Αλλά δεν μπορούν κάποιες επενδύσεις να θεωρούνται ότι είναι μονάχα στο επενδυτικό τμήμα της τράπεζας και άλλες επενδύσεις αφορούν μονάχα το τμήμα των καταθέσεων και του λιανικού τραπεζικού τομέα. Αυτό θα ήταν πολύ παράξενο. Ναι, προφανώς κυρία Πρόεδρε υπάρχουν κίνδυνοι σε όλες τις δραστηριότητες. Κίνδυνοι στις ε, λιανικού χαρακτήρα δραστηριότητες, στεγαστικά δάνεια παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό το κίνδυνο από άλλες δραστηριότητες λιανικού χαρακτήρα ή επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει αυτό να ξεχωριστεί από επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν ε, μεγάλη φερεγγιότητα. Εγώ νομίζω ότι καμία απολύτως επένδυση δεν θα πρέπει να ε, της αφαιρείται η αναγκαιότητα να καλύπτονται από τον ιδιωτικό τομέα οι απώλειες. Τώρα μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό χώρο βέβαια. Αν υπάρξει διαχωρισμός και στεγανοποίηση των κινδύνων στις τράπεζες, θα στεγανοποιηθεί και η ανάληψη κινδύνου. Εγώ νομίζω αντίθετα ότι όλοι οι μέτοχοι και όλοι οι ομολογιούχοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις, τον κίνδυνο. Αν στεγανοποιήσουμε την ανάληψη κινδύνου, φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Το πρόβλημα με τις κυπριακές τράπεζες δεν ήταν το κομμάτι των επενδύσεων των τραπεζών αυτών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι είμαι κατάπληκτος ε, που έχει τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα των καταθέσεων, γιατί αποστέλει το λαθασμένο μήνυμα προς ε, όλα τα κρατη και μπορεί ενδυνάμει να προκαλέσει πανικό. Να πω μόνο κάτι. Σε ό,τι αφορά τις απώλειες, υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα ότι ο μισθός ε, του επικεφαλής της, της ε, τράπεζας είναι 100.000 της Ιρλανδίας. Ε, την ίδια στιγμή που το κειμενόμενο επιτόκιο είναι 4,5%, το 4,6%. Άνθρωποι που είναι άνεργοι, που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και τι κάνουν οι τράπεζες, ουσιαστικά μοιράζουν τις ε, απώλειές τους και τις μετακυλίουν στους δανειολήπτε. Ενώ στην κορυφή τα πράγματα ακολουθούν την πεπατημένη. 4,6% λοιπόν είναι το κειμενόμενο επιτόκιο όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει πάνω από 100 δις ε, με ποσοστό 1%. Επομένω, το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει εμείς να πάρουμε την πλήρη ευθύνη ως πολιτική ε, ή ω υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής. Πρέπει και οι ίδιες ε, οι τράπεζες ε, να αναλάβουν την ευθύνη και να δώσουν και το καλό παράδειγμα. Θεωρούν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μοιράζουν τι απώλειέ του και να τις μετακυλίουν στους δανειολήπτε. Πρέπει πραγματικά να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στην αγορά ότι περιμένουμε καλύτερες συμπεριφορές. Εντάξει, νομίζω ότι ε, εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Συμφωνούμε όλοι μαζί σου βεβαίως. Ε, και πράγματι απαιτείται μια μεταρρύθμιση της ε, αγοράς και οι αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει την κουλτούρα και την οτροπία. Και ουσιαστικά αυτό που εμείς ζητάμε, ή τουλάχιστον αυτό που εγώ σας ζητώ, να εξετάσουμε λεπτομερώς είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα της αγοράς σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, όσοι έχουν επενδύσει λιανικού τομέα ε, να λαμβάνουν τον κίνδυνο, εγώ θεωρώ πως όχι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εμπιστοσύνη ε, στο τραπεζικό σύστημα, εκτός και αν ε, επιλύσουμε σε κάποιες από τις εγγενείς αδυναμίες ε, του συστήματος. Και βεβαίως ε, και να εξετάσω τις προτάσεις σας και τις τροπολογίες που θα καταθέσετε. Όμως νομίζω ότι με άλλους τρόπους δεν πρόκειται να έχουμε εμπιστοσύνη και θα περνάμε από κρίση σε κρίση. Γιατί στην πράξη ο υπερβολικός ε, κίνδυνος, ο πλεονάζων κίνδυνος είναι αυτός που τραβά το σύστημα προς τα κάτω. Ίσως ε, να καταλήξουμε σε κάποια διαφορετική λύση. Ίσως ε, να ακολουθήσουμε τις προτάσεις του κυρίου ε, Χόκμαρκα. Όμως, εν τέλει θεωρώ ότι είναι άδικο οι φορολογούμενοι να αναλαμβάνουν αυτό το κόστος του πλεονάζοντος κινδύνου. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Μίτσελ ότι έχω επενδύσει στην τράπεζα της Ιρλανδίας και έχασα μόνο 80% μέχρι τώρα. Εγώ είμαι μέτοχος και οπότε επομίζομαι την, το φταίξι μου. Ναι. Λοιπόν, μιλούν και δύο μιλητές μαζί. Λοιπόν, οι μέτοχοι την έχουν πατήσει πολλαπλώς, λέει κύριε. Να πάρει τηλέφωνο στο διευθυντή της, ε, της Ιρλανδίας ε, πώς δικαιολογεί ότι αυτός βγάζει 800.000 το χρόνο και 400.000 ο αντιπρόεδρος όταν ε, άνθρωποι σαν τον κύριο Σμιθ έχουν υποφέρει και έχουν τόσο μεγάλες απώλειες. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, η κυρία Μακάτη, κάθε... Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση. Α σκεφτούμε τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε Θέλω να πω ότι έχουμε προθεσμία υποβολή τροπολογιών 15 Απριλίου. Μετά θα εξετάσουμε 7 Μαΐου τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 28 Μαΐου. Θα ήθελα να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συζήτηση με τους συναδέλφους. Έχοντας ακούσει τη συζήτηση γνωρίζω ότι απομένουν κάποια ζητήματα εκρεμή που θα πρέπει να συζητηθούν εκτενέστερα. Καλώς. Θα παραδώσω την Προεδρία στο συνάδελφο Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Αιλίν. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων που θα διεξαχθεί. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Ανταλλαγή απόψεων. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολισμό 2014 ηγητής είναι ο κ. Σβέν Γκίγκολτ. Του δίνω το λόγο λοιπόν. Σβέν, έχεις το λόγο. Θα περιμένω μέχρι να μειωθεί ο θόρυβος. Ah, λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Εν συντομία, η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ για τον προϋπολογισμό του 2014 Νομίζω ότι ξέρετε ποιοι είναι οι κύριοι τομεί αρμοδιότητάς μας, είναι περιορισμένοι. Μόλον τούτο, η πρόθεσή μου είναι να ακολουθήσω την παράδοση της Επιτροπής μας στην ε, έκθεσή μου, στο σχέδιο έκθεσή μου. Θα ήθελα να ακούσω και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Για μένα είναι το να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Φορέα. Χθε καταφέραμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής της CBA, και μέσα στο νέο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας ξέρουμε ότι στο προηγούμενο σχέδιο προϋπολογισμού, στα προηγούμενα σχέδια προϋπολογισμού της Κομισιόν δεν είχαμε πάντα ε, επαρκής ε, ανταποκρίσεις στο, στις αιτήσει των τριών αυτών εποπτικών αρχών. Τους έχουμε δώσει πολλές ε, αρμοδιότητες και καθήκοντα για να δημιουργήσουν πρότυπα για τι εφαρμοστικέ και εκτελεστικέ πράξει. Αν το κάνουν αυτό όμω σε επίπεδο ποιότητα πρέπει να έχουν και την ικανότητα και του πόρου για να τα κάνουν αυτά. Αλλιώ θα έχουμε προβλήματα στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε την δυνατότητα αυτέ οι <clears throat> αποκεντρωμένε αρχέ να ανταποκριθούν στα καθήκοντά του. Το ίδιο ισχύει και για τη Eurostat και σε ό,τι αφορά την ε, διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα. Ζητούμε σε διάφορες εκθέσεις οι ευρωπαϊκές στατιστικές και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για τα φορολογικά θέματα θα πρέπει να ενισχυθεί, οπότε και εκεί πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα αυτών των φορέων για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τέλος, γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση που επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό κλάδο εδώ στις Βρυξέλλες ασκούν ιδιαίτερα ο λόμπινγκ για να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων και έχουν φυσικά την, ε, τους οικονομικούς πόρους για να το κάνουν αυτό, αλλά η κοινωνία των πολιτών δεν έχει αντίστοιχους πόρους. Έχουμε καταφέρει λοιπόν με μια παραταξιακή πρωτοβουλία να υπάρχει χρηματοδότηση για μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μπορούν να ενισχύουν το έργο τους εδώ στις Βρυξέλλες και αυτού του είδους η υποστήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν έχουμε ακολουθήσει στο παρελθόν ως της γραμμές. Πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε και τώρα αυτή την ε, πορεία και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι προτάσεις σας. Θα ήθελα να πω επίσης ότι είναι πρόθεσή μου να επισκεφθώ τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα για να συζητήσω μαζί τους το κατά πόσο τις εποπτικές αρχές μάλλον, για να δω αν είναι ικανοποιημένα, ικανοποιημένες αυτές αρχές με τον προϋπολογισμό και τη διαδικασία του προϋπολογισμού και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι ευρωβουλευτές που θέλουν να με συνοδεύσουν σε αυτές τις επισκέπτες. Αυτό θα το κάνει πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μια επίσκεψη ήδη στο Λονδίνο με τον Όλε Σμιτ. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία επισκέψεων και με τους νέους φορείς που δημιουργούνται τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σάλβα. Ε, ακολουθώ τις ε, παρενέσεις του συμβούλου μου και φίλου μου Γκοζές και θα μιλάω στα ισπανικά λοιπόν. Και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Γιάννησε που είναι η του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι εδώ, εκπροσωπούσα την Επιτροπή Προϋπολογισμών, διότι είμαι εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό 2014. Ψηφίσαμε κατευθυντήρες γραμμές, όπως γνωρίζετε την περασμένη εβδομάδα και το ψήφισμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις θα είναι ότι ε, δεν έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο ακόμα, δεν έχουμε τη νομική ε, βάση, άρα βρισκόμαστε εν κενό, ανοιχτή κατάσταση, αλλά ε, συζητήσαμε, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποβάλει πρόταση πιθανότατα από το τέλος Μαΐου που θα εδράζεται επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να πάει με κάποια πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ή κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Πρέπει να επιμείνει επί της προτάσεώς της που αποτελεί και τη βάση της προσπάθειας. Με τα χαράς άκουσα την παρέμβαση του κύριου Γκίγκολ. που αναφέρθηκε στο θέμα αυτών των ε, οργανισμών των ελευθέρων αυτών οργανισμών που είναι καθήκον της Επιτροπής ε, έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος τα τρία θεσμικά όργανα εκεί το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συναντήθηκαν έγινε μια ευγενική ανταλλαγή απόψεων περί χρονοδιαγράμματος περί εργασιών η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου ανέφερε αυτούς τους φορείς, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει πολύ στενός προϋπολογισμός για, αυτούς, για αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες, οι τρεις υπηρεσίες αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα και προσπαθούν να βρουν μια λύση για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και γι' αυτό πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι λίγο καιρού έγινε μια συνάντηση με τους τρεις αυτούς φορείς και με εκπροσώπους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, εκπροσώπους Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και έγινε μια αξιολόγηση της κατάστασης των φορέων αυτών διότι εξέφρασαν κάποια προβλήματα. Είπαν ότι εν μέρη χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εν μέρη από τα κράτη-μέλη. Και κάποια κράτη-μέλη φαίνεται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν και υπάρχει και ένα πρόβλημα ανεξαρτησίας που τίθεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους για την αντιμετώπιση της καταστάσεως. Ίσως θα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι φορείς αυτοί από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή να χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον προπολογισμό και εν μέρει από τέλη που θα καταβάλλεται από τον τομέα. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στα κράτη-μέλη. Οπότε ε, θα πρέπει να έχουμε ένα νέο σύστημα το οποίο βεβαίως θα πρέπει να είναι συμπεφωνημένο όταν συζητείται η νομική βάση για αυτούς τους φορείς. Αναφέρθηκε και ένα πρόβλημα που έχουν και θα έπρεπε να το λάβει υπόψη η Επιτροπή μας. Δηλαδή, καμιά φορά το οργανόγραμμα δεν ταιριάζει με τις ανάγκες τους. Μπορούν να έχουν αρκετά χρήματα, αλλά δεν επιτρέπεται να προσλάβουν το προσωπικό που τους χρειάζεται, διότι το οργανόγραμμα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Άρα ε, πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Εν γέννη, όσον αφορά τη διαδικασία του προπολογισμού και τις σχετικές εξέλιξεις, θα ακούσουμε την άποψη των διαφόρων επιτροπών. Θα υποβληθούν οι απόψει Επιτροπή Προπολογισμών κυρίω για προπαρασκευαστικέ δράσει και πιλωτικά προγράμματα. Έχουν γίνει προτάσεις και από αυτή την Επιτροπή. 29 Μαΐου είναι η προθεσμία για την υποβολή ιδεών. Ιδεών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μπορεί να αξιολογήσει ιδέες, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει κάποια ιδέα, αν μπορεί να την προωθήσει. Άρα να είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο το Μάιο. Η δεμή θα έλεγα ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Επιτροπή σας και άλλες ε, ειδικέ επιτροπές, καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές. Αυτό που είδαμε στους τελευταίους τρεις γύρους των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό μετά τη συνθήκη του, της Λισαβόνας είναι ότι το ε, Συμβούλιο δεν καταλαβαίνει, δεν συμμορφώνεται με το πνεύμα τη συνθήκη. Ότι είναι ισότιμη εταίροι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να εξετάσουν λεπτομέρειε. Δύο φορέ πλησιάσαμε στο να μην υπάρξει συμφωνία και να έχουμε 12, τιμόρια, αλλά πρέπει να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει με το Συμβούλιο να γίνονται σοβαρότερες συζητήσεις πιο πρώιμα. Και για να γίνει συζήτηση κάθε γραμμή, είναι ζωτικό για την διαπραγματευτική ομάδα να υπάρχει πολύ ε, στενή επαφή με τι καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές και γι' αυτό με τα χαρά παρίσταμε εδώ και θέλω να ακούσω στα όσα έχετε να πείτε. Ευχαριστώ κυρία Γένσεν. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Αρχίζω με τον κύριο Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο προπολογισμό του 2014 γιατί ξέρετε ότι εκρεμεί ακόμα το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και η νομική βάση για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Αλλά υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και θα πρέπει να είναι σαφές ότι είναι φανερό ότι θα έχουμε ένα λιτό προϋπολογισμό τα επόμενα 7 <clears throat> χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα ουσιώδη. Και η Άννε Γιάννησεν γνώριζε πολύ καλά τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα της λιτότητας αφορούν και τα προπαρασκευαστικά μέτρα και τα πιλωτικά προγράμματα. Αυτό είναι πάντα ένα από τα δικαιώματα τα οποία θέλουμε εμείς να αποκομίζουμε και να αποκτούμε από το δικαίωμα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας του προϋπολογισμού. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα τώρα στην αρχή μιας δημοσιονομικής περίοδου όταν ξέρουμε ότι σε όλα τα προγράμματα θα υπάρξουν περικοπές αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τα πιλωτικά προγράμματα υποροπαρασκευαστικές δράσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να προετοιμάσουν την σωστή εφαρμογή αυτών των ε, γενικότερων σχεδίων. Η Αν λοιπόν που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία θα ήθελα να μου εξηγήσει κατά πόσο θεωρεί ότι αυτό είναι σκόπιμο με τα πιλωτικά προγράμματα στην αρχή της δημοσιονομικής περίοδου. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι ακριβώς αυτό το θέμα των αποκεντρωμένων φορέων που όλο και περισσότερο έχουν επενδυθεί με περαιτέρω αρμοδιότητες. Έχουν πάρει δραστηριότητες για τις οποίες ουσιαστικά δεν τους δόθηκε πρόσθετο ε, προσωπικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να κόψουν το λαιμό τους εάν θέλουμε πράγματι να φέρνουν σε πέρα αυτές τις δραστηριότητες με έναν τρόπο ο είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να έχουν τις δομές και τους πόρους που είναι ε, είναι απαραίτητες για κάτι τέτοιο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στου ε, στους τριγωνικούς διαλόγους. Από τη μια μεριά δίνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δυνατότητα να έχει πρόσθετο προσωπικό και αυτό οφείλεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την εποπτική δραστηριότητα. Αλλά θα πρέπει να δούμε και με τις άλλες δραστηριότητες των αποκεντρωμένων φορέων χωρίς λοιπόν να θίξω την, την ε, ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να σκεφτούμε και τους άλλους φορείς οι οποίοι παίζουν κάποιο ρόλο σε, στα θέματα αυτά. Είδαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις των αποκεντρωμένων φορέων, είδαμε τις δηλώσεις του Τριλόγου και εμείς βέβαια δεν είμαστε μια επιτροπή η οποία διαχειρίζεται μεγάλες δαπάνες, προγράμματα μεγάλης εμβέλειας. Είμαστε περιορισμένοι λοιπόν σε ό,τι αφορά το ρόλο μας στη διαδικασία προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανάγκη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να υπάρχει μια πιο επικοδομητική προσέγγιση στη νέα δημοσιονομική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Σάλμπα. Από τους σοσιαλιστές έχει το λόγο ο κύριος Χουάν Νιόκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικροτήσω την κυρία Γιάνσεν για τα όσα είπε και για την ε, έκθεση που στήριξε την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα μας ε, στην Ολομέλεια. Επί ευκαιρία να σας συγχαρώ λοιπόν γιατί αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά φιλόδοξη για τον προπολογισμό του 2014 και απηχεί απολύτω το πνεύμα του ψηφίσματο που ψηφίστηκε στο, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από 506 βουλευτέ, όπως ξέρετε. Λοιπόν, το παρόν εγχείρημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, γιατί δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, όμως ε, με βάση την έκθεσή σας προβλέπετε και ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που φτάσουμε στο πλαφόν του 2013. Το πιο ενδιαφέρον βεβαίω είναι ότι ίσως αυτό θα επιταχύνει τη συζήτηση για τους ιδίους πόρους για το ε, επόμενο κοινοβούλιο που θα εκλεγεί του χρόνου. Εδώ λοιπόν θα ήθελα περισσότερο να αναφερθώ στα, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Οίκων που θα πρέπει να εκφέρει νομοδότηση για την διαδικασία προπολογισμού του 2014. Βεβαίω υπάρχει και η μακροοικονομική επίπτωση της ε, κοινοτική ε, ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλες οι δημόσιες δαπάνες δεν έχουν τον ίδιο μακροοικονομικό αντίκτυπο αυτό είναι σημαντικό για μας να το υπογραμμίσουμε, εφόσον πολύ συχνά υπερασπιζόμαστε τον ε, ρόλο της ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Κάποιες δαπάνες έχουν μεγαλύτερη επίπτωση από ότι άλλες. Για παράδειγμα, δαπάνες για την καινοτομία και για την έρευνα, για την ανάπτυξη. Γιατί ε, δημιουργούν προϊόν στην οικονομία, δημιουργούν ανάπτυξη στην οικονομία και οι δαπάνες ε, υποδομών που ε, προβλέπονται στη, στο τμήμα 1α της πρώτης του Συμβουλίου ε, μας μένουν πολύ λιγότερα ποσά για την καινοτομία. 15 δις για τον τίτλο 1α για 2014 βάσει του Συμβουλίου για να αυξηθεί το ποσό μέχρι το 2020 όπου θα δοθεί το δοθούν 21 δις. Είναι λίγα, δεν είναι αρκετά. Μετά, γιατί σε ό,τι αφορά την ε, μειωμένη ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και τη δέσμευση που υποθέτω ότι υπάρχει να αφοσιωθεί 3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ορίζοντα 2020. Και τώρα βρισκόμαστε περίπου στο 2%, λίγο πιο κάτω και αν έχουμε την ευελιξία που ζητάμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχουμε κάθε δυνατότητα να ε, δημιουργήσουμε μια νέα κατεύθυνση ε, των δαπανών μας προς ε, το μέλλον. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους. Ο κύριος Τόρβαλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν πολύ καλή. Δεν είμαι σε θέση να πω κάτι το οποίο να σας κάνει να ξέρετε, να γνωρίζετε περισσότερα σε αυτή τη φάση. Συμφωνώ αυτά που είπε ο κύριος Γκίγκολτ. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε μία ομάδα κρούσης, ε, θα έλεγα, για να εξετάσει περαιτέρω το θέμα. Ανάλογα με τις δυνατότητές μου θα συνεργαστώ στο βαθμό που μπορώ. Ε, αυτά μπορώ να πω για σήμερα. Ευχαριστώ. Μερσή κύριε Τόρβαλτς, ο κύριος Φίλε για την ε, Ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω την ε, κυρία Γένσεν εδώ. Συζητήσαμε στην Επιτροπή Μεταφορών για το ίδιο θέμα. Είναι πραγματικά πολύ αβέβαια τα πράγματα για τον προπολογισμό του 2014, του οποίου είναι η συγγήτρια. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ήδη λεχθέντα για τους αποκεντρωμένους φορείς. Πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα. Αν πέσουν σημαντικό ρόλο και ασκούν νέα καθήκοντα με τη νέα νομοθεσία, θα πρέπει να βρούμε τον προϋπολογισμό ο οποίος θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία αυτών των αποκεντρωμένων φορέων. Ή αλλιώ θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης εκτός του προϋπολογισμού. Από τις επιχειρήσεις ενδεχομένως τέλη τα οποία μπορούν να πληρώνουν για τις λειτουργίες που κάνουν οι αποκεντρωμένοι φορείς και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε μια τέτοια κατάσταση. Ενδεχομένω θα πρέπει να βρούμε και άλλου πόρου. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το νομικό καθεστώ των αποκεντρωμένων τομέων αλλά να μην λειτουργήσουν σωστά οι αποκεντρωμένοι φορείς ελλείψη πόρων, αυτό δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε φίλε. Και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Γκίγκολτ, εάν θέλει να κάνει κάποιο, σχόλιο. κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στα γερμανικά θα μιλήσω και εγώ και θα είμαι σύντομος. Είναι σαφές καταρχήν ότι αυτές οι... αυτή η έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα και μπορούμε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε ως Επιτροπή ΕΚΟΝ ή να περιοριστούμε στα ουσιώδη και να κοιτάξουμε μοναχά τις γραμμές του προϋπολογισμού και να έχουμε μια αντικειμενική, αν θέλετε, και επιστημονική αντιμετώπιση, αλλά ούτως ή άλλως η ίδια συζήτηση γίνεται και σε οικονομικό επίπεδο. Ξέρουμε όλοι ότι είναι σημαντικό ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεφτά των φορολογουμένων. Και εγώ ήδη ξέρω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές, ε, τουλάχιστον δύο διαφορετικές απόψεις για τα θέματα αυτά, δύο πόλοι μέσα στους οποίους θέλουμε να κινηθούμε. Και επίσης χαίρομαι και για την πρόταση που λέει ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μακροοικονομικές συνέπειες της ε, χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως σε θέματα αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι Κάτι το ιδιαίτερο όταν έρχεται από ένα Γάλλο σοσιαλιστή, αλλά και αυτό θέλουμε να το συζητήσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και μπορέσουμε επίση να συζητήσουμε ευρύτερα για το ποια θα πρέπει να είναι η λειτουργία σε μακροοικονομικό επίπεδο ενό ευρωπαϊκού προπολογισμού και επίση να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα οδηγούν σε μεγαλύτερη επανεξισορρόπηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση Ξέρουμε όμως ποιες είναι και οι ισορροπίες δυνάμεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα δεν είναι λοιπόν το ποια θα είναι τα τελικά πορίσματα, αλλά ίσως όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να βοηθήσει και τον Ευρωπαίο εκλογέα εν ώψη των ευρωεκλογών να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκονται οι διάφορες πολιτικές ομάδες για τα θέματα αυτά. Εμείς πάντως πρέπει ως Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων να αναλάβουμε τις ε, ε, ευθύνες μας και δεν πρόκειται να έχουμε ψευδεστήσεις ότι εμείς θα επηρεάσουμε τη γενικότερη συζήτηση στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου για τα επόμενα αυτά χρόνια. Απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιοι αποκεντρωμένοι ε, φορείς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Όπως είπε και ο Μάρκους, Φέρβερ, οι νομοθετικές δραστηριότητες δεν θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, αλλά πρέπει να ασκούνται από την Ευρώπη των 27. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή των άλλων αποκεντρωμένων φορών. Μέχρι τώρα είχε μονάχα ένα χαρακτήρα συντονιστικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αν υπάρξει μια συμφωνία για την CRD4, για την οδηγία κεφαλογικής απάρκειας, θα έχουμε πάρα πολλές εφαρμοστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις και αυτό σημαίνει πράγματι πρόσθετα καθήκοντα για τους αποκεντρωμένους φορείς. Και εγώ χαιρετίζω την πρόταση ότι αυτό μπορεί να καλυφθεί και από τον ιδιωτικό τομέα και όχι μοναχά από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξει μια γραμμή ε, του προϋπολογισμού η οποία θα μπορέσει να καλυφθεί με τέλη τα οποία θα εισπράττουν από τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια ξέρουμε ότι έχουμε δυσκολίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή στον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα του ενοχλεί η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερο προσωπικό για μια ευρωπαϊκή αποκεντρωμένη υπηρεσία όταν αυτά μειώνουν το προσωπικό του εθνικό επίπεδο. Αλλά εκεί πρέπει να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη ότι είναι απαραίτητε αυτέ οι δραστηριότητε από του αποκεντρωμένου φορεί. Τώρα, μια γενική συζήτηση για τα μακροοικονομικά μπορούμε να κάνουμε ούτω ή άλλω, αλλά έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα κατάλληλο προπολογισμό για αυτού του αποκεντρωμένου φορεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκίγκολτ, λέει ο πρόεδρο. Σας υπενθυμίζω ότι η κατάθεση, η παρουσίαση της έκθεσης θα είναι στις 17 Ιουνίου. 18 Ιουλίου είναι η καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες, 5 Σεπτεμβρίου η συζήτηση και ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου και η Ολομέλεια, πότε θα έρθει στην Ολομέλεια δεν το ξέρουμε ακόμα, οπότε αυτό το σημείο έχει κλείσει και μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερησίας διάταξης που είναι η συζήτηση για τις τροπολογίες της έκθεσης που αφορά το μηχανισμό παροχής οικονομικής στήριξης στα κράτη-μέλη που το νόμισμα τους δεν είναι το ευρώ. Η συγκίτρια είναι η κυρία Ντανέτα Χιούμπνερ, στην οποία δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας αναφέρω τα κύρια ε, σημεία αυτή της έκθεσης. Ενδιάμεση έκθεση που συνδέεται με τη διαδικασία της ΑΦΕΤ. Θεωρούμε όμως ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην όλη διαδικασία για τη νέα εκδοχή ε, του σχετικού κανονισμού ε, αποδέχομαι τα όσα προτείνει η Επιτροπή, ιδίως ε, την, ε, το να κινηθούμε προς ένα μεγαλύτερο φάσμα μέσων σε ό,τι φορά την οικονομική αυτή ενίσχυση. Φεύγουμε λοιπόν από την μακροοικονομική πρόληψη και πάμε σε άλλες γραμμές προπολογισμού που προσφέρουν περαιτέρω στήριξη σε αυτά τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή συνδέει αυτό τον κανονισμό με την ε, πρόσφατη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης ε, και του δημοσιονομικού και οικονομικού συντονισμού, ούτως ώστε ε, αυτό το ε, σύστημα οικονομικής ε, συνδρομής ε, να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν όμως και κάποιες προσθήκες. προς αυτόν τον κανονισμό. Θα τις αναφέρω εν συντομία. Μία από αυτές τις προτάσεις είναι ότι εφόσον θα υπάρξει, θα σταματήσει το EFSM, θα έχουμε περίπου 10 δις μη εξοποιημένης ε, ικανότητας δανειοδότησης, το οποίο θα μπορούσε να μας ε, βοηθήσει περαιτέρω, αν μπορούσαμε να εξοποιήσουμε λοιπόν αυτούς τους πόρους, ε, να το θέσουμε στη διάθεση του μέσου BOP και θα, έτσι θα αυξήσουμε την ικανότητά του από τα 50 στα 60 δις ευρώ προσθέτω επίσης ε, και πάλι στο πλαίσιο του BOP μια σύνδεση ε, με την έμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μέσω δανεισμού προς ένα κράτος μέλος. Ακριβώς με αυτό το στόχο της ε, συμβολής στην ανακεφαλοποίηση τραπεζών δεν υπάρχουν νομικές δυσκολίες. Υπάρχει λοιπόν επισήμως αυτή η δυνατότητα. Και επίσης προτείνεται όταν η συνθήκη για το ESM αλλάξει στο μέλλον να υπάρχει δυνατότητα κρατών μελών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη να ωφελούνται από την ανακεφαλοποίηση τραπεζών υπό τον ESM υπό την προϋπόθεση να ε, συμβάλλουν ε, κεφαλαιακά στο ESM. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως ε, στο πλαίσιο του ενιαίου ε, μηχανισμού εποπτείας, όπου ε, για αρκετά κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιες συστάσεις με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν. Μπορεί να υπάρξει και επικουρική δομή του e SSM για την έμεση ανακεφαλαιοποίηση και έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το επικουρικό σύστημα και στα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Μέλος του, του τμήμα του νέου κανονισμού συνδέεται και με την έκθεση Γκοζές. Η Επιτροπή προτείνει να φύγουμε από την Γκοζές και να ή μάλλον από την έκθεση Γκοζές να πάρουμε κάποια σημαντικά στοιχεία για να τα εντάξουμε σε αυτό το κανονισμό. Εγώ προτείνω όμως να αντλήσουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία από την έκθεση Γκοζές σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που συνδέονται με την ε, χρηματοοικονομική συνδρομή, την οικονομική διακυβέρνηση και την εποπτεία. Προτείνουμε λοιπόν να περάσουν περισσότερα στοιχεία από την έκθεση Γκοζέ σε αυτόν τον κανονισμό σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Δημιουργούμε και έναν ε, σύνδεσμο με την Επιτροπή Φερέιρα ιδίως για την ε, απέτηση υποβολής έκθεσης και παρακολούθησης. Υπάρχουν προτάσεις των ε, σκιωδών εισηγητών. Ε, συμφωνήσαμε όμω στα περισσότερα στοιχεία. Έχουμε καταλήξει σε συμβαστικές που καλύπτουν τα περισσότερα σημεία. Υπήρξαν ε, δύο-τρία σημεία που δεν μπορούσα να τα εντάξω σε συμβαστικέ και έτσι μένουν ω τροπολογίε. Η μία είναι η πρόταση να ε, εντάξουμε στο BOP ένα μέσο, ένα εργαλείο άμεση ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Αυτό είναι ένα μέσο που διασφαλίζεται από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να περάσουμε, να ξεπεράσουμε τα διαθέσιμα σε ό,τι φορά την ικανότητα δανειοδότησης και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ε, εκθέτει τον προπολογισμό σε άμεσο κίνδυνο. Αυτή ήταν η δική μου επιφύλαξη. Γι' αυτό εντάσσεται, ε, καταθέτεται ως ε, τροπολογία και στην έκθεση Γκοζές είχαμε και αυτή τη διάταξη που διαγράφει από την έκθεση Γκοζές. Είχαμε, έχουμε εδώ τη διάταξη μια διάταξη που συνδέει την προσβασιμότητα με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και την πολιτική συνοχής. Και πάλι εδώ έχουμε τη σύνδεση με τα διαθετικά ταμεία. Γιατί έτσι διαμορφώνεται και λειτουργεί το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Είναι κάτι λοιπόν που υπάρχει στον κανονισμό ε, πολιτικής συνοχής και διαγράφεται. Έχει διαγραφεί, δεν υπάρχει εδώ. Κάτι ακόμα που είναι αρκετά σημαντικό για μένα. Το έχουμε εξετάσει και με τον Όλι Σμιτ. Παραπομπή στο άρθρο 151 και 152 της συνθήκης, όπου έχουμε τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τη σημασία των εθνικών πρακτικών ε, στις συμβατικές ε, σχέσεις. Υπάρχει αυτός ο αυτή η παραδοσιακή σύνδεση που υπάρχει και στην ε, έκθεση Γκοσές και στα δύο αυτά άρθρα και στο άρθρο 128 της ε, Θεμελιώδους Χάρτας. Αυτή είναι, αυτό είναι το μόνο σημείο διαφωνίας που έχουμε ακόμα με τον Όλη. Να υπάρχει αυτή η αναφορά μόνο στο 152 και όχι στο 151. Κατά τα λοιπά, καταφέραμε να συνεργαστούμε με πολύ καλό τρόπο και να ενισχύσουμε το περιεχόμενο της ε, έκθεσης, ούτως ώστε να συμβάλλουμε επικοδοματικά, ελπίζουμε, στο έργο του Συμβουλίου και της Επιτροπής και πλέον η Επιτροπή και το Συμβούλιο περιμένουν την έκθεσή μας. Αν καταφέρουμε να την ψηφίσουμε τον Απρίλιο λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, να την αγνοήσει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή. Ε, συνεργαστήκαμε στενά και με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, τη νομική σκοπιμότητα κάποιων ε, λύσεων που προτείνονται. Και νομίζω ότι εν γέννη έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, αλλά με ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Κούτας από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χίμπνο για την θαυμάσια έκθεσή της και για τη συνεργασία που επέδειξε για να μπορέσουν να περιλάβει τα περισσότερα από τα σχόλια και τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει εμείς στην έκθεσή της. Για τις τροπολογίες που καταθέσαμε θα ήθελα να σταθώ στον αντίκτυπο της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις οικονομίες και τα προπολογισμού ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μιλάω εδώ για τις χώρες της Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντική η οικονομική αρρωγή προς τις χώρες αυτές για να μπορέσουν να ενισχύσουν την απορροφητική τους ικανότητα για τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι σημαντική η δυνατότητα να ενισχύσουν το φορολογικό τους, το φοροεισπρακτικό του σύστημα και να αντιμετωπίσουν την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Και επίσης να ενισχύσουμε τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις στις χώρες αυτές και την ε, εφαρμογή θεμελιωδών ανθών στην ε, Συνδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυρία Ζολή θέλει να καταθέσει αντίστοιχε τροπολογίε. Την ευχαριστούμε για τι κοινέ αυτέ τροπολογίε. Λοιπόν, υπάρχει και συνάφεια με την έκθεση του δίπτυχου του Τούπακ που έχει συγγράψει η κυρία Φερέρα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που αναφέρθηκε στο μέσο ανακεφαλαιοποίησης για χώρες που δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Το εργαλείο αυτό όμως είναι πολύ ε, καλύτερο. Αυτό θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες κύριε Λίζε. Ευχαριστώ. Ο Όλη Σμίτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Την ευγνωμοσύνη μου εκφράζω προ την Τανούτα Χούμπνερ. Είναι πάντα προνόμιο να συνεργαστεί κανείς μαζί σου. Ε, ναι, ε, Όπω τα βλέπω, τα πράγματα είναι σημαντικό νομοθέτημα αυτό ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Και έχουμε την πρόκληση όσον αφορά τις διαιρέσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή να αντιμετωπιστεί. Έχουμε τις χώρες που είναι εντός και τις χώρες που είναι εκτός. Σημερίζομαι τις απόψεις σου ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, μικρές διαφορές, αφορά την ε, αιρεσιμότητα, το έχουμε θέσει ξανά, καταλαβαίνει τα επιχειρήματά μας. Απ' την άλλη κατανοούμε και αυτό που λες δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εδώ. Καταλαβαίνω όμως την προσέγγιση σου τελικά. Αναφέρθηκε στο άρθρο 151 και 51-52. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις για τη διαμόρφωση των μισθών και των αμοιβών και πώς οι κοινωνικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη στα κράτη-μέλη. Και ήταν άλλο ένα από τα σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν για την αποδοχή του six-pack, διότι υπονομευόταν το όλο σύστημα Κάποιος θα το έλεγε σκανδιναβικό, βόρειο μοντέλο ή οτιδήποτε. Μοιραζόμαστε την ευθύνη. Δεν εξαρτάται από τους πολιτικούς η διαμόρφωση των μισθών και των ημερημιστίων, ακόμα και των ελαχίστων αυτών. Όπως τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Το θέμα είναι ζωτική σημασίας. θεωρούμε ότι χρειάζεται ξεχωριστή ψηφοφορία. Άλλοι ίσως να μην το θεωρούν τόσο σημαντικό το ζήτημα. Πολιτικός όμως, πως για τον επιμερισμό των ευθυνών για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, στη χώρα μου τουλάχιστον, αυτό είναι σημαντικό θέμα. Εν γέννη, σε ευχαριστώ. Πολύ καλή προετοιμασία για την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα αργότερα σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Σμιθ για τους πρασίνους. Η κυρία Ζολή έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χούμπνερ έξοχη η έκθεσή της. Θέλω να της πω ότι η ομάδα μου είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την έκθεση ως έχει σήμερα. Θα υποστηρίξουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες και θέλω να ποτίσω φόρο τιμής στο πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε η κυρία Χούμπνερ και κατέστησε έτσι δυνατή την επεξεργασία του κειμένου. Παραμένουν δύο θέματα που θα θέλαμε να αναφέρονται εκτενέστερα, να πηγαίνουν πιο μακριά. Η διατύπωση της συμβαστικής F θα θέλαμε να είναι πιο ισχυρή όσον αφορά τη δυνατότητα ανακεφαλοποίησης, άμεσης ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, αλλά μπορούμε να δεχτούμε το μηχανισμό ως τον περιγράφει η κυρία Χιούμπνερ. Δεν κατανοώ γιατί συστήνει αρνητική ψηφοφορία για την τροπολογία με παριθμόν 53 δεν είναι τίποτα παρά κείμενο που αναπλάνεται από την έκθεση Γκοζές και αναφέρεται στην εξής δυνατότητα όταν υπάρχει απόκληση σε σχέση με το πρόγραμμα προσαρμογής μιας χώρας, να, άρα είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση της χώρας, θέλαμε να μπορεί να γίνει επαλήθευση κατά πώς αυτή η απόκληση οφειλόταν στο ίδιο το πρόγραμμα προσαρμογής ως είχε ψηφιστεί το κείμενο, ως το έχω συμπεριλάβει στην έκθεση Γκοζές. Πέραν αυτών, εγώ και η ομάδα μου είμαστε υπέρ της ομάδας και θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ κυρία Ιωλή. Από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Φίλε. Χωρίς μικρόφωνο, ο μιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χούμπνερ Είχαμε πολλές συναντήσεις ε, μεταξύ των συντονιστών και είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την αυριανή ψηφοφορία. Μερικά σχόλια τα οποία για μένα είναι σημαντικά. Καταρχήν η συμβαστική τροπολογία C που αφορά την ε, μεταφορά από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης στο Μηχανισμό Υποστήριξης του Ισοζυγίου Πληρωμών, του BOP και επίσης συμβαστικές τροπολογίες E και F για την έμεση και άμεση επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Εγώ χαίρομαι που παραμένουμε στην προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος, του ESM. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί πλήρως σε νομικό επίπεδο, αλλά είναι σωστή κατεύθυνση να μπορέσει και για τις χώρες αυτές να ακολουθηθεί ο δρόμος της, ε, ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσα στα πλαίσια του ESM με την υποστήριξη των ισοζύγιων πληρωμών ως υποκατηγορία. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτήν την ε, προσέγγιση που θα πρέπει να αφήσει τις αλλαγές στα διαρθρωτικά ταμεία να γίνουν μες στον κανονισμό των διαρθρωτικών ταμείων και όχι στο τρέχον νομοθέτημα. Είναι πολύ καλή έκθεση. Δανούτ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε φίλε. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Χούμπνερ, εάν θέλει να παρέμβει. Πιθανότατα δεν έχω πολλά να προσθέσω. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια μέρα χωρίς να καταλάβουμε γιατί μπορούμε να αναφερθούμε και στα δύο άρθρα. Διότι γι' αυτό το έκανα. Ήθελα να αναφερθώ και στα δύο, και στο 151 και στο 152 και εσύ επιμένει στο ένα. Και μα λες ότι διαφέρουμε πάνω σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όμω θε να έχει αναφορά μόνο σε ένα άρθρο δηλαδή μόνο κοινωνική εταίρη... χωρί ε, συμβατικέ σημασιακέ διευθετήσει. Θυμάμαι τι συζητήσει με του Ιδού συναδέλφου στα πλαίσια του ΣΥΚΣΠΑΚ, όπου το άρθρο 151 ήταν εξίσου σημαντικό για αυτού. Αλλά εν γέννη, κατά τα άλλα, συμφωνούμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συζητητές για τις συζητήσεις, διότι έμαθα πολλά και εγώ και ήταν εξαιρετική η όλη διαδικασία. Βέβαια και εγώ ίδια θα είμαι κατά της άμεσης ανακεφαλοποίησης επί τη βάση του μέσου αυτού όπου υπάρχει άμεση σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Γι' αυτός, και αυτός είναι ο μόνος λόγος, διότι από τις συζητήσεις που είχα με τους εμπειρογνώμονες κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποια όρια σχετικά με το τι μπορούμε να πάρουμε από τις χρηματοστικές αγορές, από τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Με την εγγύηση από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ότι υπάρχουν όρια και κυρίως αν θέλει να το κάνει κανείς αυτό για την, άμεση, για την, έμεση, ανακεφ, για την άμεση ανακεφαλοποίηση όπου εκθέτει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό στους κινδύνους που πάντα συνδέονται με τη λειτουργία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Αυτός ο κίνδυνος πιθανότατα είναι πάρα πολύ ψηλός. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, αυτός είναι ο πρακτικός λόγος για τον οποίο είμαι κατά της άμεσης ανακεφαλοποίησης. Αλλά κατανοώ ότι ήταν μια αρχή που έπρεπε να έχουμε αυτά τα μέσα, αυτός στόχο που θα επιτρέπουν την άμεση ανακεφαλαιοποίηση και γι' αυτό το αναφέρω εδώ, αναφέρω αυτή την ιδέα. Δηλαδή το ESM να είναι επικουρικής μορφής. Δηλαδή για να μειώνεται η άμεση σχέση μεταξύ ενός ε, θεσμού όπως είναι το ESM και των χρηματοστικών ιδρυμάτων που θα γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση τους μέσω των ταμείων. Αυτή είναι η προσωπική αμφιβολία που έχω και γι' αυτό δεν προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το BOP για την άμεση ανακεφαλοποίηση. Δεν είμαι κατά της άμεσης ανακεφαλοποίησης αυτής καθ' αλλά κατά της χρήσεως του BOP, δηλαδή του κανονισμού για τον ε, ισολογισμό των πληρωμών, ισορροπία των πληρωμών. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Χίμπνερ. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έγγελ. Ευχαριστώ πρόεδρε, μπορώ να είμαι σύντομο. σύντομα λοιπόν και εμείς χαιρετίζουμε το έργο της ε, κυρίας Φίμπνερ και των σκιωδών εισηγητών. Ε, η Επιτροπή δεσμεύεται να ενσωματώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα αποτελέσματα της συζήτησης ε, αυτής της έκθεσης και να λάβει υπόψη και το σχετικό κομμάτι της έκθεσης Φερέρ, αν και εκεί ήταν λίγο διαφορετική ε, η περίπτωση. Το γνωρίζετε αυτό. Και ξέρετε ότι δεν έχουν επικυρώσει ε, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο όλα τα κράτη-μέλη που δεν ε, συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε το Συμβούλιο να εντάξει αυτό το μέσο στην εργαλειοθήκη. Είναι μια καλή ιδέα για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Ε, συμμεριζόμαστε τις ε, επιφυλάξεις της συζητήτριας για την σκοπιμότητα ένταξης αυτού του μέσου ε, στην εργαλειοθήκη γιατί θα μας εκθέσει σε ενδεχόμενες απώλειες. Σημειώνουμε τα υπόθηκαν για το ESM. Ξέρουμε ότι είναι βέβαια αρμοδιότητα των κρατομελών, δεν μπορώ να πω πολλά από αυτού. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την αναφορά στα 151 και 152, τα, αυτά τα δύο άρθρα, έχω δύο παρατηρήσεις. <clears throat> Πρώτον, η συνθήκη Ισχύει, όπω και να έχει. Είτε γίνεται η παραπομπή, είτε όχι. Πρέπει να εφαρμόζονται τα άρθρα, όπως και να έχει. Και μετά, όσοι συμμετείχατε στην εξέταση της έκθεσης γοζες ε, θα θυμάστε ότι ε, ε, οι διατυπώσεις ε, επιλέχθηκαν πολύ προσεκτικά. Επομένω, μπορούμε να τη στηρίξουμε αν ε, ακολουθήσουμε αυτή τη διατύπωση. Αν ξεφύγετε από αυτή, τότε θα υπάρχουν ουσιαστικέ δυσκολίε. Ευχαριστώ κύριε Άγγελ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Χούμπνερ, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλο του σημείου αυτού. Σα υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, στην αυριανή πρωινή συνεδρίαση και μία τώρα ανακοίνωση πριν κλείσουμε το απόγευμα θα έχουμε ένα μονάχα σημείο στην ημερήσια διάταξη στις 4.30 γιατί στις 3 θα λάβει χώρα η ανοιχτή συνέλευση των Προέδρων. Το σημείο στην για διάταξη θα είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη ορισμένων δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά την, ε, πληροφο... την... Ε, τις πληροφορίες των δημοσιονομικό ή τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον λογιστικό έλεγχο και έχουμε φτάσει στο τέλος της συνεδρίας. Ευχαριστώ όλους και όλες.